Dear colleagues, let's start. Uh, I submit to you uh, the following changes to the draft agenda. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην ημερησία διάταξη. Έχουμε ένα νέο επτά για την uh, διαφραμένο διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης το διορθωτικό ε, για το ίδιο Λάιζα της κυρίας Μακοβέη αναβάλλεται για τις ανθρωπιστικού τύπου χορηγήσεις θεωρήσεων αναβάλλεται επίσης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις με αυτές τις τροποποιήσεις θεωρούνται δεκτές. 11 Ιουνίου τώρα του 18 συνεδρίαση 2 Ιουλίου του 18 παρακαλώ να εγκρίνετε τα πρακτικά υπάρχουν καθυστερήσεις στις μεταφράσεις των πρακτικών θα σας υποβληθούν στις επόμενες συνεδριάσεις Ξεκινάμε λοιπόν την αποκοινού συζήτηση με την Επιτροπή δημοσιονομικού ελέγχου. Σας καλωσορίζω συνάδελφοι. δημιουργήθηκε η θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στα πλαίσια της ενισχυμένης συνεργασίας. Η νομική βάση παραμένει το άρθρο 86 της συνθήκης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να μας δώσει περισσότερα στοιχεία ενημέρωσης. Ε, οι αρμοδιότητες ε, ε, από πλευράς μας περιορίζονται σε περιπτώσεις απατών εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα πρέπει να υπάρχει μια συνενετική διαδικασία για την θέση στη λειτουργία του EPPO χωρίς ε, να υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με τα μέσα τα οποία είναι υποδιαπραγμάτευση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά από την ε, προπαρασκευαστική φάση των τριών ετών θα τεθεί σε λειτουργία πλήρως το EPPO από το τέλος του 2020. Ως εκ τούτου τα εφαρμοστικά μέτρα για την επιλογή και λειτουργία <clears throat> του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και του Σώματος των Ευρωπαίων Επιμέρους Εισαγγελέων έχει ήδη ξεκινήσει και γι' αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ορίσει τον κύριο Αντώνιο Μούρα Ιταλό Εισαγγελέα ως εκπρόσωπό του. Ε, στόχος της Επιτροπής Ελέγχου και Επιλογής θα είναι η δημιουργία ενός ε, συνοπτικού καταλόγου υποψηφίων και η αξιολόγηση των ε, ικανοτήτων και των προσόντων των υποψηφίων. Έχουν τεθεί αρκετές ερωτήσεις σχετικές με τις εφαρμοστικές προϋποθέσεις για τη θέση του βασικού εισαγγελέα σε σχέση με την ηλικία του και τη διάρκεια της εντολής, αυτά θα συζητηθούν. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να πω ε, στον κύριο Τάραντα μήπως θέλει να κάνει μία μικρή εισαγωγή. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας μέρα. Είναι δύσκολο για μένα να αντικαταστήσω την κυρία Γκρέσλε η οποία είναι πολύ δύσκολη στην αντικατάστασή της αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις εκ μέρους της παρακαλώ. Εμείς θεωρούμε ότι είναι θετική η ευκαιρία που μας δίδεται να ανταλλάξουμε απόψεις για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα σε σχέση με την υπηρεσία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Θα θέλαμε επίσης να σας ανακαινώσουμε ότι προχωρά η επεξεργασία του κειμένου από πλευρά της αρμόδιας κοινοβουλευτική επιτροπής σε σχέση με τη στελέχωση της υπηρεσία αυτής και ε, θα ενημερωθούμε ως προς αυτό γραπτά σύντομα. Ο λόγος είναι ότι εκφράστηκαν κάποιες ανησυχίες από τις συμμετέχουσες ε, χώρες ε, σχετικά με το ε, ιδιαίτερα χαμηλών φιλοδοξιών αν θέλετε χρονοδιάγραμμα το οποίο θα οδηγήσει στη λειτουργία του γραφείου του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα. Αυτό ε, δυσκολεύτηκε ακόμα περισσότερο Υπάρχουν δύο χώρες επιπλέον και αυτό σημαίνει ότι λιγότερα ε, ε, πόροι θα είναι διαθέσιμοι από κάθε χώρα. Αυτά θα πρέπει να συζητηθούν σε μια άλλη κοινή συνάντηση σε λίγες εβδομάδες με την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να σας μεταφέρω εκ μέρους της κυρίας Γκρέσλετ σήμερα. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σόνκα από την Αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω έρθει εδώ, έχει έρθει και η κυρία Χόφμαν από την υπηρεσία Όλαφ και θα πάρουμε ένα αλλάξ τον λόγο. Θα ήθελα να πω το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε σχέση με τις συζητήσεις για την εφαρμογή των αποφάσεων μέχρι τώρα από πλευρά των κρατών μελών και η κυρία Χόφμαν θα σας δώσει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με το δημοσιονομικό κομμάτι. Όπως πολύ σωστά υπογραμμίσατε σήμερα το πρωί, Πρόεδρε, στην εισαγωγή σας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπλέκεται με δύο τρόπους. Πρώτον, δίδοντας κατευθυντήριες γραμμές μέσω των ψηφισμάτων του και μέσω του διορισμού του κυρίου Μούρα στην Επιτροπή Επιλογής που θα οδηγήσει στην δημιουργία του συνοπτικού καταλόγου των υποψηφίων και την αξιολόγηση των συγκεκριμένων υποψηφίων. Για να διευκολυνθεί η διαδικασία έχει ξεκινήσει και μια νομοθετική διαδικασία στο Συμβούλιο σχετικά με, τις προτάσεις, ε, με θέμα τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 13ης Ιουλίου υιοθετήθηκαν από το αρμόδιο πάνελ του Συμβουλίου οι λεγόμενοι κανόνες λειτουργίας όπως ακριβώς και είχαν προταθεί από πλευράς μας. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή για μια ακόμη φορά ενέκρινε μια δεύτερη σειρά προτάσεων την 31η Ιουλίου για μια άλλη εφαρμοστική απόφαση από πλευρά του Συμβουλίου για τον διορισμό των μελών της Επιτροπής Επιλογής. Πρόκειται για ένα κατάλογο ο οποίος περιλαμβάνει 12 μέλη που περιλαμβάνει και το μέλος το οποίο έχετε προτείνει εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον κύριο Μούρα. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο θα υιοθετήσει την εφαρμοστική του απόφαση ή απόφαση απλή του Συμβουλίου, θα δούμε πώς θα είναι, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου έτσι ώστε να ξεκινήσει τις εργασίες επιλογής η ομάδα αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Κάποια στιγμή το μήνα Νοέμβριο ελπίζουμε. Ο κανονισμός ε, ε, προβλέπει να δημιουργηθεί όπως είπαμε από την Επιτροπή αυτή ένα συνοπτικός κατάλογος υποψηφίων και περιλαμβάνει επίσης και μια τεκμηριωμένη ε, γνωμοδότηση σχετικά με τις ικανότητες και τα προσόντα των υποψηφίων. Ε, φυσικά γι' αυτό θα πρέπει, αυτού μάλλον θα πρέπει να προηγηθεί ε, η κήρυξη χειρεύουσας θέσης. Αυτό έχει ήδη γίνει μέχρι τώρα. Το Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο θα οδηγήσει στον διορισμό, είναι αρμόδια επί του διορισμού αρχή και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νομίζουμε ότι η κήρυξη χειρεύουσας θέσης θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα ήδη κατά τη διάρκεια του ε, Σεπτεμβρίου γιατί περνάει ο καιρός και θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο διορισμός τον Μάρτιο του 19. Αυτό σημαίνει ότι εσείς σαν κοινοβούλιο πριν τις επόμενες εκλογές θα κληθείτε να πάρετε μια απόφαση. Ταυτόχρονα συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της ομάδας εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε ορίσει τις συγκεκριμένες απαιτήσει που υπάρχουν για τη θέση του Ευρωπαίου Ισαγγελέα. Αυτό δεν είναι ε, κήρυξη χειρεύουσα θέση, είναι μια περιγραφή των απαιτήσεων για τη συγκεκριμένη θέση. Ε, περιγράφει ακριβώς αυτά τα οποία θα θέλαμε να δούμε όταν δηλώσουν τους υποψηφίους τους ε, τα κράτη-μέλη. Πρέπει να στείλουν τρία ονόματα σύντομα έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής. Και τέλος θα ήθελα να πω ότι για τα θέματα προσωπικού εμείς έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες κήρυξης ενδιαφέροντος για τις θέσεις που θα χρειαστούν και για την Έχουμε προχωρήσει σε διευθετήσεις και για την ψηφιακή πλατφόρμα. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι υπεύθυνη έως ότου το EPPO εν πάση περιπτώσει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού λειτουργίας του έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με εκπροσώπους των συμμετεχουσών χωρών. Είναι 22 οι χώρες αυτές μέχρι σήμερα όπως είπα υπήρξαν δύο επιπλέον από τις τελευταίες εβδομάδες. Μέχρι τώρα έχουν γίνει τρεις συναντήσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων και η τέταρτη θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα. Ασχολούμεθα στα πλαίσια της ομάδας αυτής με θέματα εφαρμοστικού τύπου και θα αναφερθούμε επίσης την επόμενη εβδομάδα στα μέτρα τα οποία έχουν λάβει τα κράτη-μέλη από πλευρά τους έτσι ώστε να εντάξουν στις νομικές τους αρχιτεκτονικές την θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Η διαδικασία θα κρατήσει όπως ξέρετε δύο χρόνια έτσι ώστε όλοι να είναι έτοιμοι την ίδια στιγμή. Για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες των κρατών μελών δημιουργήσαμε επίσης και μια ψηφιακή πλατφόρμα. Στα πλαίσια αυτής της πλατφόρμας μπορούν να ανταλλάξουν πληροφορίες νομικής φύσεως ή και απλές ενημερώσεις μεταξύ τους και έχουμε δώσει διάφορες κατευθυντήριες γραμμές. Πρόκειται για μια διαδραστική πλατφόρμα η οποία διευκολύνει την επικοινωνία και την εφαρμογή των ε, αποφάσεων που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα. Θα ήθελα να ζητήσω από την παρακαθήμενή μου να συνεχίσει με τα υπόλοιπα θέματα. Σε ευχαριστώ Πίτερ. Και σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμπληρώσω τα όσα είπε ο, Πίτερ με κάποια ακόμα στοιχεία προς ενημέρωσή σας σε σχέση με αυτή την ε, έκθεση και συζήτηση με τα κράτη-μέλη για το πώς να εφαρμόσουμε τη τις διάφορες ε, πτυχές ε, κεφάλαια μάλλον αυτού του συστήματος θα γνωρίζετε ότι ένα στοιχείο ήταν η οδηγία που συζητήθηκε στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ όπου τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να μεταγράψουν σε εθνικό νόμο μέχρι τον Ιούλιο του επόμενου έτους. Η προθεσμία είναι σχετικά σύντομη και αυτή η οδηγία αφορά την προσέγγιση των ε, δικημάτων που αφορούν τον ευρωπαϊκό ε, προπολογισμό και πρέπει να μεταγραφεί στο ποινικό δίκαιο των κρατών μελών. Ένα σημαντικό στοιχείο για την εργασία του Ευρωπαίου ε, εισαγγελέα, γιατί ακριβώς αφορά τις αρμοδιότητες του μελλοντικού Ευρωπαίου εισαγγελέα και του γραφείου του, του επιτελείου του. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πού βρίσκεται η μεταγραφή της οδηγίας στα κράτη-μέλη και πάλι η προθεσμία είναι πολύ σύντομη και πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε καλύτερα να ολοκληρώσουμε αυτές τις προσπάθειες. Ο κύριος Στάραντ ανέφερε ε, τον προϋπολογισμό του γραφείου του Ισαγγελέα Γνωρίζετε ότι το σχέδιο προπολογισμού του 2019 υιοθετήθηκε από την Κομισιόν το Μάιο. Η πρόταση περιλαμβάνει μέχρι στιγμής ένα σύνολο πιστώσεων 4,9 εκατομμύρια για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί η πρόσληψη προσωπικού. Ξεκινάμε με το 2019 με τον επικεφαλή και φυσικά, επικεφαλής και φυσικά με τους Ευρωπαίους ε, εισαγγελείς και 1,9 εκατομμύρια προβλέπονται για την ανάπτυξη ε, για το, του συστήματος διαχείρισης των ε, υποθέσεων του Ευρωπαϊκού του Γραφείου Εισαγγελικού Γραφείου. Η Ολλανδία και η Μάλτα προσχώρησαν ε, στο σύστημα ε, και είμαστε ευτυχείς που έγινε αυτό. Αλλά φυσικά ε, χρειάζεται και περισσότερο προσωπικό λόγω αυτής της εξέλιξης. Λαμβάνουμε υπόψη φυσικά την ανακοίνωσή σας ότι Λίμπε και Κόντ θα στείλουν κοινή επιστολή στην Επιτροπή για τον προϋπολογισμό και την στελέχωση και φυσικά θα λάβουμε υπόψη την επιστολή σας και τα αιτήματά σας ε, τώρα. Η Κομισιόν συνεργάζεται με τις αρχές του Λουξεμβούργου έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια ε, σωστή έδρα για το Ευρωπαϊκό, τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα. Έχουμε προχωρήσει θετικά. Ίσως να γνωρίζετε ότι οι αρχές του Λουξεμβούργου προσέφεραν δωρεάν ένα ε, κτίριο που βρίσκεται κοντά στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι ο πύργος Β, έτσι είναι γνωστό. Ε, και ε, αυτή τη στιγμή συζητάμε σε τεχνικό επίπεδο ώστε να αξιολογήσουμε τις λειτουργικές ανάγκες του ΕΠΟ για να μπορέσει να λειτουργήσει, όπως είπαμε, σωστά. Είναι τεχνικές οι συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Τέλος, θα ήθελα επίσης να αναφέρω. Είμαι και Διευθύντρια Πολιτικής της Όλαφ και γνωρίζω πολύ καλά ότι οι Ευρωπαίοι Εισαγγελές και οι Όλαφ θα πρέπει να συνεργαστούν στενά στο μέλλον. Αυτό περιλαμβάνεται και στον κανονισμό για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα και η Κομισιόν ανέλαβε να αναθεωρήσει τον κανονισμό περί Όλαφ ώστε να ε, συντονιστεί με τις διατάξεις για τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα να συμπεριληφθούν λοιπόν εκεί οι απαραίτητε διατάξεις που θα ευνοήσουν την ε, αγαστή συνεργασία ανάμεσα στο ΕΠΟ και στην ΟΛΑΦ. Η Κομισιόν προτείνει και διάφορες σκόπιμες αλλαγές ώστε οι έρευνες της Όλαφ να γίνουν ακόμα πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές. Προσβλέπουμε στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο ε, για αυτή την πρόταση. Όπως γνωρίζετε, ο χρόνος τρέχει και η Κομισιόν θα ήταν ευτυχής αν οι συνομοθέτες το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα μπορούσαν να έρθουν σε ε, συνεργασία πριν από τις ε, χειμερινέ διακοπέ. Προσβλέπουμε, όπω σα είπα, σε στενή συνεργασία με το Κοινοβουλίο. Ωραία, σα ευχαριστώ πολύ. Πριν να δώσω το λόγο στα μέλη για ερωτήσει και παρεμβάσει, θα ήθελα να σα υποβάλω εγώ κάποιε ερωτήσει για τι ε, πόρου ε, για το προσωπικό. Ο προπολογισμό που έχει προβλεφθεί, σα φαίνεται αρκετό. Η Κομισιόν πώ προχώρησε για, στην αξιολόγησή τη, η Κομισιόν χρησιμοποίησε την προεκβολή για να λάβει υπόψη και τα νέα κράτη-μέλη που ζήτησαν συνεργασία για, όσον αφορά την ε, πρόσληψη προσωπικού. Σύμφωνα με το άρθρο το οποίο θεσπίζει το ΕΠΠΟ, η Κομισιόν μπορεί να ορίσει μετά από διαβούλευση με το Συμβούλιο έναν, ε, έναν ε, υπάλληλο της Κομισιόν ώστε να λειτουργήσει ως διοικητικός, ε, ως διοικητής, ως διευθυντής μάλλον. Η Κομισιόν έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχει δηλαδή ένας προσωρινός διευθυντής που έχει οριστεί, διοριστεί. Όσον αφορά τον διορισμό του Ευρωπαίου Επικεφαλής Εισαγγελέα, Ποια είναι η διαδικασία για να συμμορφωθούμε προς το άρθρο 14. Έχει η Κομισιόν προετοιμάσει την πρότασή της όσον αφορά το σχήμα επιλογής, την οργάνωση τώρα του εισεργασίας του ΙΠΠΟ. Σύμφωνα με το άρθρο 21, η διοργάνωση του εισεργασίας του ΙΠΠΟ θα διέπεται από το εσωτερικό κανονισμό και η Ευρωπαίος ε, επικεφαλής της εισαγγελίας ε, θα ε, υποβάλει πρόταση για την, τον εσωτερικό κανονισμό που θα πρέπει να υιοθετηθεί από το σύνολο των εισαγγελίων. Ωστόσο, ο εισαγγελέας θα πρέπει να μην ξεκινήσει από το μηδέν. Έχετε προετοιμάσει λοιπόν ένα σχέδιο και αν ναι, τα κράτη-μέλη έχουν συνδεθεί με αυτή την εργασία πώς θα ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Κρίνσπεκ από την ε, ε, ΛΥΜΠΕ. Έχουμε όμως το συνήθειο στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, ο καθένας να παίρνει το λόγο για δύο λεπτά, σας θυμίζω. Merci, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομη. Με τους συναδέλφους ε, και εγώ χαίρομαι για την πρόοδο αυτού του ε, φρακέλου που ε, βρισκόταν μέσα στις προθέσεις της Ευρωπαϊκής εδώ και πολλά χρόνια. Χαίρομαι λοιπόν για την οργάνωση και για τις πληροφορίες που μας δώσατε και θα είμαι σύντομη λοιπόν να σας ευχαριστήσω. Το ερώτημά μου είναι άμεσο. Είμαστε πολλοί και στην κοινοβουλευτική μου ομάδα που ζητάμε πώς θα μπορούσε να προβλεφθεί η επέκταση των αρμοδιοτήτων για ε, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Πέρυσι, στον οδικό χάρτη που επέβαλε, παρουσίασε μάλλον ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ανακοίνωσε τη δημοσίευση μιας ανακοίνωσης για μια πιθανή επέκταση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία σε σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που αποτελεί για όλα τα κράτη-μέλη ένα από τα κύρια θέματα ανησυχίας τη κοινή γνώμη όσον αφορά την ασφάλεια. Θα μου απαντήσετε ίσως πως θα υπάρξει ομιλία την επόμενη εβδομάδα για την κατάσταση της Ένωσης, αλλά ε, εκμεταλλεύομαι τη ε, παρουσία σας για να σας ρωτήσω τι γίνεται με αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κλίντ. Σήμερα Έχω κοντά μου δύο παιδιά μου και τέσσερα εγγόνια. Για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες. Ήρθαν να δουν πώς εργαζόμαστε. Θα συνεχίσω στα γερμανικά τώρα, αφού αυτά σας τα είπα στα αγγλικά. Φορέστε τα ακουστικά σας. Η σημερινή υπόθεση είναι πολύ σημαντική, ιδίω όταν σκέπτομαι τι μου λένε οι ψηφοφόροι μου. Κυρίως εννοώ το οργανωμένο έγκλημα και όχι μόνο για τα φορολογικά θέματα, αλλά βεβαίως και τα λεγόμενα εικονικά νομίσματα τελευταία. Για την επόμενη δημοσιονομική προοπτική βλέπουμε ότι θα χρειαστεί να αγωνιστούμε και για το τελευταίο ευρώ που θα χρειαστούμε για να εκτελέσουμε εδώ τα καθήκοντά μας, δηλαδή ε, της χρηματοδοτής ευρωπαϊκής ε, πολιτικής. Χαίρομαι λοιπόν που δημιουργείται τώρα καθιδρύεται ο θεσμό τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να μπορέσουμε επιτέλου να επιτύχουμε κάποιε πρόοδου. Εκφράζω ρητά τη λύπη μου για το γεγονό ότι δεν συμμετέχουν όλε οι χώρε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν συμμετείχαν όλε, θα είχαμε την ευκαιρία να ενισχύσουμε από την αρχή και βεβαίω να διευκολύνουμε τη συνεργασία μεταξύ Όλαφ και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να μπει σε μια πιο υγιή βάση. Τώρα η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων είναι κάτι που θα πρέπει να προκύψει από δύσκολες διαδικασίες στο μέλλον. Δεν είναι δεδομένη. Πράγματα που ίσως η όλα αυτά θεωρήσει ότι είναι διοικητικά παραπτώματα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ίσως να τα θεωρήσει ήδη αξιόπινα αδικήματα. Θα χρειαστεί λοιπόν πολύ προσοχή. Δίστανται οι απόψεις βέβαια για τα θέματα αυτά, αλλά είμαι πεπισμένος ότι εάν δεν χάσουμε το στόχο από τα μάτια μας θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πρόοδο. Πολύ σημαντικό είναι το θέμα της ΕΠΟ, διότι βεβαίως από την άλλη μεριά οι πολίτες έχουν κουραστεί να βλέπουν να δημιουργούνται διαρκώς νέοι θεσμοί. Η δε κριτική αντιμετώπιση και επικριτική αντιμετώπιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αυξηθεί. Θα το δούμε αυτό και στι επόμενε ευρωεκλογέ. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξεκαθαριστεί στους πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα των πολιτών, των ψηφοφόρων και φορολογουμένων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριο Τάραντ. Ο κύριο Τέρι Κάμπρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, στα αγγλικά. Εγώ έχω συντάξει πέντε ερωτήσεις εδώ. Όμως ορισμένες καλύφθηκαν, μένουν μόνο δύο. Δεδομένων των ενδεχομένων συνδέσμων μεταξύ εκτελεστικής εξουσίας και εισαγγελέων σε ορισμένες χώρες μέλη. Πώς θα εξασφαλίσουν οι χώρες μέλη την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υπό διπλή κεφαλή. Δεύτερο, ποιες είναι οι προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ό,τι αφορά τις μη συμμετέχουσε χώρες. Ε, θυμίζω το σχόλιο που μόλις έκανε ο κύριος Κλίντς. Δύο λοιπόν ε, ξεκάθαρες αλλά σύντομες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κ. Στάραντ. Ο κ. Λόπεθ Αγγιλάρ. Uh, Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι κάτι το οποίο θα σημαδέψει αυτήν την κοινοβουλευτική περίοδο και επίσης και την περίοδο της συγκεκριμένη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο βασικός ρόλος δεν είναι δικός μας, δεν είναι μια τακτή νομική διαδικασία, αλλά έχουμε εμπλακεί στην διαδικασία αυτή καθ' όλη τη διάρκεια τους Συνεπώς λοιπόν έχουν υπάρξει πολλά στοιχεία τα οποία συζητήθηκαν μέχρι τώρα. Τώρα έχει φτάσει η στιγμή να αξιολογήσουμε σωστά την στρατηγική εφαρμογής των συγκεκριμένων ρυθμίσεων και γι' αυτό ακριβώς απαιτείται αρκετή συνεργασία ανάμεσα στην ίδια την ΕΠΟ ε, και στα κράτη-μέλη, σωστή συνεργασία και ταυτόχρονα απαιτείται να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι και συγκεκριμένες προτεραιότητες γύρω από την επίτευξη των στόχων οι οποίοι δικαιολογούν αν θέλετε και τεκμηριώνουν την ύπαρξη της υπηρεσίας αυτής. πολέμηση εναντίον των απατών, καταπολέμηση των απατών εν πάση περιπτώσει, των φορολογικών απατών, που επηρεάζουν ε, τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Εγώ ήμουν εισηγητής ε, για την οδηγία η οποία αναφέρεται στην προστασία ε, των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσω ποινικών διαδικασιών. Και γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να γνωρίζουμε λίγο καλύτερα για τη διάρθρωση των εργασιών της ΕΠΟ, οι οποίες θα πρέπει να διασφαλίζουν πλήρως τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. ιδιαίτερα σε περιπτώσεις απατών εις βάρος του κοινοτικού προϋπολογισμού και μάλιστα για μεγάλα ποσά μερικές φορές. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να εκτιμήσουμε ε, το μέγεθος των απατών αυτών. Συνολικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι εντός και εκτός της Ένωσης χάνονται 50 δις ε, της βάση. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται να κάνουμε βήματα προοδού για την προστασία της Ένωσης από τα οικονομικά αυτά εγκλήματα. οι προσπάθειες πρέπει να γίνουν και από την Ένωση και από τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια ουσιαστική αξιολόγηση της κατάστασης και χάραξη της στρατηγικής την οποία θα ακολουθήσει ε, η υπηρεσία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. κυριακή Κινίτσι ένα, η τελευταία ομιλήτρια. Δύο λεπτά παρακαλώ. Εμείς σαν φιλελεύθεροι μπορούμε να μιλάμε όσο θέλουμε, αλλά η πρακτική εδώ είναι τα δύο λεπτά για να απαντήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους ε, διαδοχικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΟΛΑΦ σχετικά με τη θέση σε λειτουργία της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. και εμένω στην επιστολή που έστειλε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, στην οποία είμαι αναπληρωτή, έτσι ώστε να υπάρξουν κάποιες απαντήσεις ε, γύρω από την ανάγκη πλήρους κάλυψης και προστασίας των ευρωπαϊκών οικονομικών συμφερόντων. Ε, βέβαια εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες, όχι μόνο η ΟΛΑΦ αλλά και η Europol όπως επίσης και η Eurojust. Πώς λοιπόν θα πετύχουμε τον στόχο αυτό. Ε, ποιες διαδικασίες προβλέπετε να ακολουθηθούν και όχι μόνο διαδικασίες αλλά ποιοι είναι και οι ανθρώπινοι πόροι ε, οι οποίοι θα απαιτηθούν για να παίξει σωστά τον ρόλο της η Europol. Τώρα ε, σχετικά με τις δύο χώρες οι οποίες θα συνεργαστούν, αυτό διευρύνει την ενισχυμένη συνεργασία, αλλά θα ήθελα να μάθω ε, με ποιες δράσεις, με ποιο τρόπο και με ποιους πόρους η Όλαφ θα μπορέσει να διευκολύνει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην περίπτωση διεθνικών έρευνων σε χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν στην συγκεκριμένη υπηρεσία της εισαγγελία. Ελπίζω να σεβάστηκα τα δύο λεπτά, λέει η κυρία Κινίτσι. Θα ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει και συνοπτικά και ελπίζω με γραπτό τρόπο να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις. Θα απαντήσω σε κάποιες από αυτές και μετά ο Πίτερ Τζόνκα θα συμπληρώσει ε, τις απαντήσεις. Και φυσικά αν έχετε γραπτέ ερωτήσεις ε, θα σας απαντήσουμε. Επανέρχομαι στο θέμα που σας απασχολεί πολύ, δηλαδή τους πόρους για τη, ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. Ρωτήσατε αν είναι παρκής η Κομισιόν έκανε πρόταση για τον προϋπολογισμό του 2019 που είναι υποσυζήτηση, υποδιαπραγμάτευση με τη Δημοσιονομική Αρχή, τις Δημοσιονομικές Αρχές, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και φυσικά είναι πρόθεση και επιθυμία της Κομισιόν ε, Θα δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από τις διαπραγματεύσεις και όπως είπα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την σύναψη, μάλλον την συμμετοχή των δύο χωρών, Μάλτα και κάτω χώρες. Ολλανδία. Θα ήθελα επίσης να πω, αναφέρατε και ήδη ακούστηκε για την ε, ε, προσωρινή, ε, τον προσωρινό διευθυντή, διοικητικό διευθυντή, ναι, η Κομισιόν έχει σχεδόν ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Κάτι άλλο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι ε, είπε ο κύριος Τάραντ μισό λεπτό ο κύριος Κάμπρας το είπε ναι, σε σχέση με τους ε, εισαγγελείς ε, των κρατών μελών οι κανόνες είναι ξαφείς μέσα στον κανονισμό του ΕΠΟ και όταν ενεργούν για το ΕΠΟ να είναι ανεξάρτητοι και να είναι ε, υπό την αρμοδιότητες και υπό την ε, ε, διέπονται από τους κανόνες της ΕΠΟ. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να κάνουμε να και να στελεχώσουμε το σύστημα για, μέσω του συστήματος των αποσπασμένων εισαγγελέων. Η κυρία Κινίτσι ανέφερε και τη συνεργασία με τη Europol και άλλους οργανισμούς και αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση για το μέλλον γιατί έχουμε διάφορους φορείς σε αυτό το τομέα Europol, Eurojust και τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε την συνεργασία ανάμεσα στις ε, οργανισμούς διευθυντής ε, θα δει τον διευθυντή της Europol μέσα στο Σεπτέμβριο ώστε να ξεκινήσει και καλά η συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς τους δύο οργανισμούς. Ε, νομίζω και ο κύριος Κλίνς ε, συμφωνεί. Είναι κρίμα που όλα τα κράτη-μέλη δεν είναι εκεί. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι εύκολο να στελεχωθούν πλήρως τα δύο αυτά σώματα, ε, αλλά νομίζω πως η Κομισιόν έχει ενισχύσει τον κανονισμό της όλα ώστε να μπορέσει να υπάρξει ομαλή συνεργασία. Βεβαίως πάντοτε θα πρέπει να υπάρχει η βούληση Θέλουμε λοιπόν η συνεργασία αυτή να είναι ισχυρότερη και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε ολόκληρη την Ένωση. Αυτή είναι η επιθυμία μας και δίνω το λόγο στον Πίτερ. Ευχαριστώ Μαργαρέτα. Προφανώς δεν είμαι η κυρία Σρόντερ, όπως λέει εδώ μπροστά η ταμπέλα. Είναι, είμαι ο Πίτερ Σόγκα. Ε, θέλω λοιπόν να συμπληρώσω τα όσα είπε η Μαργαρέτα. Καταρχάς, για την υπόθεση των αποσπασμένων εισαγγελέων. Υπάρχει ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο που ορίζει το καθεστώς των αποσπασμένων εισαγγελέων. Ακόμα και αν έχουν διπλή θέση πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και υπάρχουν διαδικαστικές και ε, ε, διαδικασίες για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία. Δηλαδή μπορεί μια υπόθεση να αφαιρεθεί ε, από τον εισαγγελέα. Αν υπάρξουν υπόνοιες ότι δεν είναι ανεξάρτητος και θα υπάρχουν και ασφαλιστικές δικλείδες στον εσωτερικό κανονισμό για τον τρόπο με τον οποίο πληρώνεται ο άνθρωπος αυτός, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος όταν εργάζεται σε ευρωπαϊκά θέμα, για ευρωπαϊκά ζητήματα. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι αυτός, αυτή η σύνδεση που ανέφερε ο κ. Κάμπρας ανάμεσα ε, στην Εθνική Εισαγγελία και την Ευρωπαϊκή δεν θα είναι ε, δεν θα επηρεάζει. Γιατί ακριβώ είναι η ραχοκοκαλιά του ΕΠΟ. Για την ερώτηση του κύριου Λόπε Αγγιγιάρ, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργήσει αποτελεσματικά στα κράτη-μέλη. Όντω, πολλά διακυβεύονται εδώ. Εμείς ε, έχουμε με τα κράτη-μέλη από την πρώτη μέρα της πρακτικής εφαρμογή έχουμε συνεργαστεί μαζί του συχνά για τα, το τι πρέπει να γίνει. Ε, ακολουθούμε την ε, διαδικασία εφαρμογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο και θα εξασφαλίσουμε ότι αφιερώνουν επαρκή χρόνο και πόρους για να εφαρμόσουν την νομοθεσία και για να ορίσουν τους σωστούς ανθρώπους. Ε, πρώτον ως υποψήφιους για το Ευρωπαίους Εισαγγελείς και δεύτερον για τους Ευρωπαίους απεσταλμένου εισαγγελείς. Και τώρα, για να απαντήσω στην κυρία Γκρινσμπέκ ε, για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ε, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για θέματα τρομοκρατίας. Όντως, είναι προτεραιότητα για κάποια ε, κράτη-μέλη. Η Κομισιόν έχει προβλέψει και μέσα στην ομιλία του κυρίου Γιούνκερ πέρυσι αναφέρθηκε μια ανακοίνωση με προοπτική το 2025. Αυτή η ανακοίνωση θα βγει την επόμενη εβδομάδα. Θα, θα, θα δημοσιευτεί την επόμενη εβδομάδα και προβλέπεται μεταρρύθμιση του σημερινού πλαισίου για την καταπολέμηση της συνοριακής τρομοκρατίας στα κατημέλη μας με μια σειρά θεμάτων που τονίζουμε και όπου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα μπορούσε να ε, ε δείξει την αξία της, ε, αποδεικνύει γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η σωστή μέθοδος για να απαντήσουμε σε αυτού του είδους τη δημοκρατία; ε, τώρα, για τις χώρες που δεν συμμετέχουν. Μένουν έξι κράτη-μέλη και προσεχώς μπορεί να είναι και πέντε που θα μείνουν ε, έξω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και πρέπει με αυτό να εργαστούμε. Έχουμε έναν μηχανισμό συνεργασίας περίπλοκο, ειδικά στο κανονισμό για το την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ε, και βέβαια και μέσω της στήριξη της Όλαφ και οι μηχανισμοί εκτό της Ευρωπαϊκής Αγγελία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ε, συμμετέχουν τα κράτη-μέλη. τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναγνωρίζουν ε, την ειλικρινή συνεργασία που είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούν με αυτό και να αναγνωρίσουμε τις οδηγίες, τις, τα συντάλματα, ε, τα εντάλματα συγγνώμη, τα οποία ε, θα εκδίδει η εισαγγελία, ε, να αναγνωρίζουν τη δικαστική συνεργασία και αλληλοβοήθεια. Ελπίζουμε λοιπόν πως σύντομα θα έχουμε το νομικό πλαίσιο με τα κρατημέλη. Ήδη υπάρχουν οι βάσεις στον κανονισμό για την εισαγγελία. Ορισμένα κρατημέλη θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο. Θα δούμε πώς θα το διοργανώσουμε αυτό αλλά έχουμε μια επαρκή βάση μέσα στον ίδιο τον κανονισμό για να το κάνουμε. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα ζητήσω από τον κύριο Νίμαερ από την Προεδρία του Συμβουλίου αν θέλει να χρησιμοποιήσει ε, και να πάρει το λόγο για λίγο. Α, κυρία Νίμαερ. Σας καλωσορίζουμε όλους. Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία είναι υπό εξέταση στο Συμβούλιο στην παρούσα φάση. Καταρχήν η κήρυξη ε, για την ε, κενή θέση του εισαγγελέα που θα οδηγήσει σε ιστερότερη φάση στο διορισμό. Οι υποψήφοι θα πρέπει να ολοκληρώσουν θητεία 7 ετών που δεν θα ανανεούνται και ε, θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψουν την θητεία τους αυτή πριν φτάσουν στην ηλικία της συνταξιοδότησης και όχι πάνω από 70 ετών. Αυτό περιλαμβάνεται στην τελική απόφαση σχετικά με το διορισμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Θα πρέπει να αποδεχθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την, το υπόμνημα σχετικά με την κήρυξη σε χειρία της συγκεκριμένη θέση είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την ανεξαρτησία του Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε στο Συμβούλιο. Ε, το δεύτερο θέμα είναι η Επιτροπή Επιλογής Ήδη κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών και πριν από τις διακοπές και μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τα πράγματα προχώρησαν αρκετά καλά. Στις 12 Σεπτεμβρίου στο Κορεπέρ θα τα συζητήσουμε. και μετά μπορεί να τεθεί πλέον σε εφαρμογή η σωστή λειτουργία του συγκεκριμένου πάνελ από το μήνα Οκτώβριο. Σας ευχαριστώ. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί σήμερα το απόγευμα και σε επίπεδο συντονιστών και όπως είπε και η κυρία Γκροστέτ ε, θα υπάρξει μια από κοινού επιστολή των δύο επιτροπών. Σας ευχαριστώ για την συμπροεδρία. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, τον Ιούνιο του 18, στις 18 Ιουνίου υπήρξε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα, ε, τα διαχειριστικά συμβούλια των, ε, ε, της, που θα λειτουργήσουν στα πλαίσια των πολιτικών αποφάσεων για την μετανάστευση και την υποδοχή προσφύγων. Σήμερα λοιπόν συγκεντρωθούμε σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης όπως επίσης και στη διαχείριση των λεγόμενων ολοκληρωμένων μορφών εξωτερικών συνόρων. Υπάρχει και μια γνωμοδότηση η οποία θα πρέπει να συζητηθεί σαν τμήμα αυτής της γενικότερης συζήτησης σχετικά με τον τεχνικό εξοπλισμό ο οποίος θα είναι απαραίτητος. Υπάρχουν εκπρόσωποι λοιπόν των equipment ε, fund are reporters for these files. Ε, Mr. Francesco Gazzello Όλοι αυτοί οι ομιλητές λοιπόν θα μας παρουσιάσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων μέσων όπως προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά θα είναι σε θέση να δώσουν απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Ξεκινάμε με τον πρώτο ομιλητή. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να παρουσιάσω την υπηρεσία μου. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και θα είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Σας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Πάρα πολύ σύντομα για τα επόμενα Έχουμε κάποια εμπειρία σε σχέση με τις αξιολογήσεις τις οποίες έχουμε ήδη κάνει και τις οποίες έχουμε ήδη παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Ταμείο. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να εκμεταλλευτούμε τα μαθήματα από το παρελθόν αυτών και να μην επαναλάβουμε τα λάθη τα οποία είχαμε κάνει όπως την έλλειξη ευελιξίας, την έλλειξη σωστού συντονισμού, απαιτείται επίσης περισσότερη απλούστευση, απλοποίηση αν θέλετε και θα πρέπει να έχουμε συστήματα τα οποία να είναι πλήρως κατανοητά στα κράτη-μέλη. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε την έλλειψη ευελιξίας που είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Εμείς προχωρήσαμε στην κατανομή των ποσών για το 2014 με αριθμούς του 2012 αλλά όταν η κρίση κορυφώθηκε σε σχέση με μετανάστες και με ε, πρόσφυγες το 15 2016 τα χρήματα δόθηκαν σε λάθος χώρες. Δηλαδή τα στατιστικά τα οποία είχαμε στοιχεία ήταν από το 10, 11, 12 και 13. Αυτό δεν αντικατόπτριζε την κατάσταση το 14 και το 2015. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και όταν παίρνουν τις πιστώσεις αυτές τα κράτη-μέλη θα πρέπει αμέσως να ανταχορηγούν καλύπτοντας συγκεκριμένες προτεραιότητες τις οποίες έχουν. Νομίζω ότι απλά θα μάθουμε όπως είπα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν. Τώρα βλέπουμε την κατανομή του προϋπολογισμού. Βλέπετε εδώ το, στα πράσινα ε, το ταμείο ε, για το άσυλο 10 περίπου δις μια μεγάλη αύξηση σε σχέση με το ισχύον δηλαδή μιλάμε για τριπλασιασμό περίπου για τη διαχείριση των συνόρων έχουμε 8 δις είναι ε, κάτι και αυτό πολύ ανώτερο από προηγούμενα χρόνια Τώρα για τις εξωτερικές υπηρεσίες. ...860 εκατομμύρια και για την υπηρεσία Frontex και την υπηρεσία για τη διαχείριση των συνόρων ε, θα προβλέψουμε περίπου 12 δις σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους. Τα πράγματα είναι παρόμοια με αυτό το οποίο είχαμε κάνει στο παρελθόν. Καταρχάς, πρέπει από κοινού να έχουμε ένα ευρωπαϊκό εναρμονισμένο σύστημα χορήγησης ασύλου, το οποίο να στηρίζει την νόμιμη μετανάστευση προς τα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να δοθούν εγγυήσεις στους νόμιζους μετανάστες ε, και ταυτόχρονα να αντιμετωπιστεί και να καταπολεμηθεί η, ε, μη νόμιμη, οι μη νόμιμες μορφές ε, μετανάστευσης. Πώς θα το κάνουμε αυτό τώρα. Καταρχάς έχουμε πολύ συγκεκριμένα μέσα όπως κίνητρα για επανεγκαταστάσεις και μεταφορές επίσης υποψηφίων για, διεθνή προστασία. Ενισχύουμε επίσης τις εθελοντικές επιστροφές. Καλύπτουμε επίσης τις ανάγκες των υποχρεωτικών επαναπροωθήσεων. Βελτιώνουμε τις διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Ένα άλλο σημαντικό θέμα και δεν είναι μια απλή δήλωση από πλευράς Επιτροπής για καλύτερη μορφέ συντονισμού. Απλά προσπαθούμε η μετανάστευση, η ένταξη ε, των μεταναστών να συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα μέσα τα οποία πολλές φορές έχουν πολύ, περισσότερα, πολύ περισσότερες οικονομικές δυνατότητες από τα επιμέρους μέσα τα οποία είμαστε σε θέση να χρησιμοποιούμε. Επίσης και εξωτερικά μέσα τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία έχουν συζητηθεί σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο για τη μετανάστευση και τον έλεγχο των συνόρων. Στην ουσία προσημιούνται κάποιες πιστώσεις έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά τα οποία υπάρχουν λόγω της μη επάρκειας των υπαρχουσών οικονομικών δυνατοτήτων. Παρά την αύξηση λοιπόν των ποσών, παρά την εγγυήσει που έχουμε για την αύξηση των ποσών για το άσυλο και τη μετανάστευση, θα υπάρξει και πρόβλεψη στο νέο αυτό ταμείο έτσι ώστε ε, κάποιες ε, δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν για συγκεκριμένες δράσεις ε, να μπορούν να ε, εφαρμόζονται και να διεξάγονται και σε τρίτες χώρες και όχι μόνο στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. η ερώτηση από πλευρά των εμπλεκομένων είναι ότι αν πράγματι ε, το κοινωνικό ταμείο μπορεί να βοηθήσει σε θέματα ένταξης των μεταναστών πώς ε, θα μπορέσετε να συνδυάσετε τα μέσα αυτά με τα δικά σας μέσα χωρίς να δημιουργηθεί σύγχυση. Εμείς έχουμε κάνει κάποιους διαχωρισμούς ανάλογα με τη φύση των διαστηριοτήτων και δεν είναι θέμα χρονοδιαγράμματος. Καταρχάς, ε, ε, εμείς με το δικό μας ταμείο θα μπορέσουμε να δράσουμε στην πρώτη φάση, σε ό,τι είναι απαραίτητο στην αρχή της διαδικασίας. Τα πρώτα μέσα δηλαδή, τα οποία θα απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν για να καλυφθούν οι ανάγκες ε, των μεταναστών. Αυτό θα κρατήσει ίσως έξι μήνες, ένα χρόνο, όχι ένα μήνα βέβαια, αλλά είναι η φύση αυτής της δραστηριότητας όπως η εκμάθηση βασικών στοιχείων της γλώσσας υποδοχής. Όλα αυτά είναι μέσα τα οποία θα βοηθήσουν επίσης και στην πρόσβαση ε, στην αγορά εργασίας η οποία όμως θα στηριχθεί στην δεύτερη φάση από το κοινωνικό ταμείο. δεν θα χρησιμοποιήσουμε το κοινωνικό ταμείο άμεσα για τα μέτρα υποδοχής σαν παράδειγμα των μεταναστών. Απαιτείται λοιπόν εδώ προσπάθεια για να αποφύγουμε επικαλύψεις σε ορισμένους τομείς. Έχουμε κάνει λοιπόν προσπάθειες έτσι ώστε να διευκρινίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα υποστηρίξουμε συγκεκριμένες δραστηριότητες. θα προσπαθήσουμε οι εξωτερικές υπηρεσίες της Ένωσης να παίξουν ρόλο ακόμα μεγαλύτερο σε σχέση με την καταγραφή της ε, συγκυρίας κάθε φορά. Και με το συγκεκριμένο οικονομικό μέσο διασφαλίζουμε αρκετά μεγάλη ευελιξία μόνο το 50% θα δίδεται στα κράτη-μέλη στην αρχή της προγραμματικής περίοδου το 10% θα δίδεται ε, μετά το 2024 και το 40% θα δίδεται ανατριετία καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου για τη στήριξη των νέων προτεραιοτήτων. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο φιλόδοξοι από ό,τι μέχρι τώρα Επαναλαμβάνω ότι το 40% θα χορηγείται σε τριετή βάση. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε ε, να καλύψουμε αυτά τα προβλήματα στα οποία αναφέρθηκα πριν, να είμαστε ε, προσαρμοστικοί, ε, να μπορέσουμε να καλύψουμε τις τοπικές ανάγκες σε σχέση με τα στοιχεία τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας την επόμενη τριετία. Τώρα για το ολοκληρωμένο Ταμείο Διαχείρισης Συνόρων. Αυτό είναι ένα επιπλέον μέσο που θα επιτρέπει ε, και τελωνιακούς ελέγχους και τον έλεγχο των προσώπων τα οποία είναι υπομετακίνηση. Θα πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων όπως επίσης και την πολιτική στον τομέα των θεωρήσεων. Εδώ βλέπετε τον εξοπλισμό που έχουμε ανάγκη, δηλαδή σκάφη, ελικόπτερα, συστήματα εκπαίδευσης, ηλεκτρονικά συστήματα, διαλειτουργικότητα και εξυγχρονισμός των μέσων άσκησης της πολιτικής αυτή. Συνεργασία λοιπόν ε, με και με τις ε, ε, υπηρεσίες ελέγχου των εξωτερικών συνόρων είναι κάτι το απαραίτητο. Από τη μία έχουμε την υπηρεσία και από την άλλη έχουμε τα κράτη-μέλη. Εμείς δεν χρηματοδοτούμε την ίδια την υπηρεσία, αλλά χρηματοδοτούμε τα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Απαιτείται λοιπόν συνεργασία ανάμεσα στην υπηρεσία αυτή και τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών, τις αρχές των κρατών μελών. Τώρα για τα συστήματα πληροφορικής τα οποία χρησιμοποιούνται έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τίθεται το θέμα της χρηματοδότησης των πληροφορικών συστημάτων σε εθνικό επίπεδο και σε συγκεντρωτικό επίπεδο μέσω του EU -LISA. Ενώ τα εθνικά συστήματα θα χρηματοδοτούνται με, δικά μας, με δικές μας πιστώσεις. Επίσης κάποια θέματα θα καλύπτονται το κόστος τους από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Λοιπόν, αυτά δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα, να πω ότι εμείς και στον τομέα των θεωρήσεων και της διαχείρισης των συνόρων κάνουμε το ίδιο όπως και πριν, 50% στην αρχή της προγραμματικής περίοδου με βάση τις στατιστικές 18, 19 και 20. Θα δίνουμε επίσης το 10% από το 24 και μετά με βάση τα στοιχεία τα οποία θα έχουμε το 22 και 23 και το 40% οι λεγόμενες θεματολογικές διευκολύνσεις θα δίδονται ε, σε ετήσια ή διετή βάση έτσι ώστε να καλυφθούν επίγουσες ανάγκες. Ε. Τελειώνει, τελειώνει. Τώρα πρώτη, προτινόμενες βελτιώσεις ε, στα, ναι, σε αυτά καταπιστεύματα ή ταμεία μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη ευελιξία, περισσότερες προϋποθέσεις ε, για την χρήση τους, λειτουργική στήριξη βελτιωμένη ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε και τις απαιτούμενες διορθώσεις. Θα δίδονται ε, επίσης, θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης ορισμένων πιστώσεων όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Επίσης ε, θα ζητείται η επιστροφή πιστώσεων όταν διαπιστωθεί η μη χρήση τους. Υπάρχουν ε, θέματα και ε, ε, προγράμματα όπως το AMF τα οποία υποστηρίζονται κατά 10% ιδιαίτερα σε επίπεδο λειτουργικών συστημάτων πληροφορικής και θα πρέπει να υπάρξει σωστός παραλληλισμός με την λειτουργία άλλων μέσων σύμφωνα με τον κανονισμό ο οποίος είναι σε ισχύ και θα τελειώσω με αυτό, θα προτείνουμε επίσης και ένα υψηλό επίπεδο συγχρηματοδότησης για κάποια θέματα τα οποία παρουσιάζουν υψηλή προσ... Ε, ε, υψηλό ενδιαφέρον. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους προτείνουμε τις ε, λεγόμενες αν θεματικές ή θεματολογικές παρεμβάσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το σύνολο των κοινωτικών προτεραιοτήτων με ευέλικτη χρήση των διαθέσιμων πιστώσεων. Λοιπόν, η απλοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Το θέμα είναι πώς θα αυξήσουμε την απλοποίηση μέσω της αναθεώρησης των εθνικών προγραμμάτων Θα έχουμε επίσης επιλογές κόστους οι οποίες θα απλοποιηθούν και αξιολογούνται ταχύτερα. Εδώ βλέπετε τα μέσα με τα οποία αντιμετωπίζουμε τα θέματα της μετανάστευσης. Κοιτάξτε, θα πρέπει να τελειώσετε κύριε Περιμένουμε λοιπόν τον Επίτροπο Κίνγκ στις 10. Παρακαλώ λοιπόν ολοκληρώστε τα όσα είχατε να πείτε. Μάλιστα. Α, τελειώσατε. Ωραία. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Περολάτ, γιατί θα μας παρουσιάσει την πρότασή της. Έχετε δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη για να πω ότι έχουμε προτείνει μια, ένα τελείως ε, νέο ολοκληρωμένο ταμείο, κονδύλι, ταμείο για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των κρατών μελών για τη χρηματοδότηση ε, του εξοπλισμού ε, τελωνιακού ελέγχου, που ελέγχουν δηλαδή τα αγαθά που περνάνε από τα εξωτερικά σύνορα. Ένα τέτοιο ξεχωριστό ταμείο ε, διαφορετικό από το Customs One είναι ότι μπορεί να λάβει υπόψη την έλλειψη ισορροπίας στην ε, εκτέλεση των συνοριακών ελέγχων, των τελωνιακών ελέγχων μάλλον ανάμεσα στα κράτη-μέλη που καταλήγουν όχι μόνο σε διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη αλλά και λόγω διαφορετικών ε, δυνατοτήτων και πόρων ε, θέλουμε να συμβάλλουμε στους ελέγχους μέσω μιας σωστής ε, χρηματοδότησης του ελεγκτικού εξοπλισμού και έτσι να μην υπάρχει διαφορετική ροή των ε, αγαθών προς τη πιο αδύναμα σημεία των συνόρων. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το δεύτερο σκέλος του ολοκληρωμένου ταμείου χρηματοδότησης των συνόρων. Ε, έχω μόνο δύο διαφάνειες, γι' αυτό θα είμαι πολύ σύντομη. Ε, θα βάλουμε μόνο στην ε, διαφάνεια στα διάφορα πράγματα ώστε να μπορέσω γρήγορα να σας τα παρουσιάσω. Ο γενικός στόχος αυτού του κονδυλίου 1,3 δις είναι για 7 χρόνια να στηρίξουμε, είναι να στηρίξουμε την ε, Τελωνιακή Ένωση ώστε να εξασφαλιστούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και των κρατομελών, να αυξήσουμε την ασφάλεια και να υπάρξει συντονισμός, ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνονται οι νόμιμες ε, ε, επιχειρηματικές δραστηριότητες. Θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε την αγορά, διατήρηση και αναβάθμιση αξιόπιστων ε, ε, εξοπλισμών ε, τελωνιακού ελέγχου. Μιλάμε δηλαδή για μη παρεμβατικούς εξοπλισμούς όπως η ακτίνες Χ, τα αυτόματα συστήματα σκάν, κινητά, κινητές συσκευές και αυτό δεν έχει να κάνει με τα όσα σας παρουσίασε ο Φρανσίσκο υπό την διαχείριση των θεωρήσεων. Δεν θα χρηματοδοτήσουμε IT. Ε, Αυτό θα χρηματοδοτηθεί από, το, ε, από άλλα προγράμματα. Θα είναι μόνο για κρατημέλη, δεν θα είναι για υποψήφιες χώρες, ούτε για άλλες, καμία άλλη χώρα και για να χορηγηθούν αυτά τα χρήματα θα προχωρήσουμε πρώτα σε μια αξιολόγηση των αναγκών από τα κράτη-μέλη ανάλογα με το είδος των συνόρων και μέσω της επιτροπολογίας θα θεσπίσουμε προγράμματα εργασίας για να χορηγηθούν αντίστοιχα και τα κονδύλια. Η αξιολόγηση των αναγκών θα είναι πολύ σημαντική γιατί έτσι θα χορηγήσουμε τα κονδύλια ανάλογα με το είδος των συνόρων και σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε μια αξιολόγηση των αναγκών για κάθε είδος ε, συνόρου γιατί το κάθε είδος συνόρου είναι διαφορετικό και χρειάζεται διαφορετικό εξοπλισμό. Πρέπει να γίνει ε, αξιολόγηση χερσαία πήγε, ε, μάλλον χερσαία ε, αέρια κτλ. Ε, τελευταία μου διαφάνεια είναι αυτή όπου μπορώ να σας εξηγήσω τις σχέσεις ανάμεσα στον εξοπλισμό ελέγχου που πάλι αφορά μόνο για την αγορά ε, συγκεκριμένων ε, ε, τεχνολογιών και του προγράμματος ελέγχου των τελωνίων, αξιολόγηση αναγκών, κατευθύνεις γραμμές, κατάρτιση και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Και εδώ σταματώ. Ευχαριστώ. Thank like... Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ασφαλώς, η γραμματεία μας θα διανύμει τις PowerPoint παρουσιάσει που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα μέλη τη Επιτροπή μα. Ευχαριστώ τον ε, Επίτροπο κύριο Κίνγκ για την έλευσή του, τον καλωσορίζω. Θα ακούσουμε μόνο τους συζητητές, η κυρία Ντάλη πρώτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα λάβω το λόγο εξ ονόματος της κυρίας και εξ ονόματος της κυρίας Τάνια Φαγιών θα αρχίσω με το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης για το οποίο είμαι συγγήτρια που πιστεύουμε ότι είναι ένα μέσον που θα μας επιτρέψει να βρούμε τρόπους να στηρίξουμε τις χώρες μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη μετανάστευση και πρόσωπα που ζητούν άσυλο, χρηματοδότηση 10 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ πριν ήταν μόνο 2. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει στις χώρες μέλη και στην Ένωση να εκπληρώσουν τις υποχρώσεις τους. Είναι σημαντικό να μην χαθεί ο βασικός στόχος, δηλαδή της αλληλεγγύης. Έχω λοιπόν κάποιες ερωτήσεις προς τον κύριο Επίτροπο. Πρώτα, αλληλεγγύη ως στόχος. Πολύ σημαντικός. Ωστόσο, θέλω να μάθω από την Επιτροπή γιατί η αρχή της αλληλεγγύης δεν αποτελεί πλέον πρωταρχικό στόχο του Ταμείου. Για άλλο θέμα τώρα, μπορεί ο Επίτροπος να εξηγήσει περισσότερο πώς θα διασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση για κάθε ένα από τους στόχους του Ταμείου σε κάθε χώρα μέλος και δεν θα πρέπει να υπολογίσουμε ένα ελάχιστο ποσοστό για κάθε ένα από τους στόχους για τη δράση του Ταμείου εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πηγαίνουν χρήματα σε άλλες χώρες, ενώ υπάρχουν από το IMF δηλαδή, από το Ταμείο δηλαδή Ασύλου και μετανάστευση, ενώ υπάρχουν και άλλες πηγές. Για τους co-performance indicators, αυτή είναι ποσοτική. Δεν θα πρέπει η Επιτροπή να επιλέξει μάλλον μια ποιοτική προσέγγιση, για παράδειγμα απασχόληση, ε, παιδιά των μεταναστών στα σχολεία και ούτω καθεξής. και θα παρακολουθεί τη χρηματοδότηση των έργων και την εκτέλεσή τους και θα ενημερώνει το Κοινοβούλιο. Θα προχωρήσω βεβαίως σε στενή συνεργασία με όλους τους συζητητές και σκιώδεις συζητητές και αν μου επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε θα πω τώρα αυτά που έχει σημειώσει εδώ η Τάνια φαγιών. Η κυρία Φαγιών είναι κολλείεται σήμερα Γι' αυτό θέτω ερωτήσεις στον Επίτροπο εκ μέρους της. Και εγώ και η κυρία Φαγιών θεωρούμε ότι τα χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία είναι πολύ σημαντικά για την Ένωση και για τους πολίτες της για να μεταφερθούν σε, στην πραγματικότητα, σε πραγματικές δράσεις οι χρηματοδοτήσεις αυτές και να διασφαλιστεί ότι οι δράσεις αυτές απηχούν το τι αναμένουν οι πολίτες από εμάς τους πολιτικούς. Έχοντας υπόψη τα διάφορα εργαλεία εξωτερικής πολιτικής εξωτερικών δράσεων, ρωτώ τον Επίτροπο, γιατί η Επιτροπή προτίθεται να χρηματοδοτήσει δράσεις σε τρίτες χώρες που σκοστοχεύουν σε εσωτερικές πολιτικές. Πρόκειται για οριζόντιο θέμα, το οποίο μπαίνει και στο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Επί της ουσίας, η ρωτά ποιος είναι ο ρόλος των παραρτημάτων και γιατί δεν περιλαμβάνονται στο κυρίως σώμα του κανονισμού. Επίσης, δείκτες, πεδίο εφαρμογής και άλλα θα έπρεπε να περιλαμβάνονται. Σε ό,τι αφορά τους στόχους των κανονισμών, οι δράσεις που θα πρέπει να περιλαμβάνονται θα πρέπει να είναι και της συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής. Από την άλλη μεριά αυτά δεν απηχούνται πλήρως στις προβλέψεις. Και ρωτά γιατί η κυρία Φαγιών και δεν θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο ποσοστό το οποίο θα, χρηματοδοτείται, το οποίο θα προβλέπεται μάλλον για τη χρηματοδότηση του κάθε στόχου. Τελευταία δε ερώτηση, έχοντας ακούσει από ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ότι υπάρχουν δύο μέρη, δύο τμήματα μάλλον τα οποία τους απασχολούν, αύξηση δηλαδή της διαφάνειας της χρηματοδότησης κλπ. Πολλές ερωτήσεις βέβαια, αλλά ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας δώσει κάποιες πρώτες απαντήσεις. Αλλά και γραπτός αργότερα. Ευχαριστώ πολύ, Λέναρτς. Δύο θέματα. Πρώτα, το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Όπως η προλαλήσασα, χαίρομαι διότι η νέα πρόταση ενισχύει τον προϋπολογισμό του Ταμείου και δείχνει ότι αυτό είναι σημαντικό και για το προσεχές μέλλον της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης. Διεξάγονται αυτές οι λεπτομερείς συζητήσεις τώρα παρόλο που δεν έχουμε ακόμα σημειώσει καμιά πρόοδο διότι είναι ανοιχτά όλα τα ντοσιέ ασύλου και μετανάστευσης. Σωστό είναι και το Συμβούλιο να προχωρήσει και να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις μαζί μας. Η ερώτησή μου επίσης είναι γιατί δεν θεωρεί πλέον την αλληλεγγύη ω πρωταρχικό στόχο του Ταμείου, αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών μελών. Σε ό,τι αφορά την κατανομή, είναι σημαντικό που βλέπουμε ότι η καταπολέμηση παράνομη μετανάστευση και οι επιστροφέ παίζουν τώρα σημαντικότερο ρόλο, διότι θεωρώ ότι είναι ο πιο αδύναμο κρίκο σε όλη την αλυσίδα τη πολιτική μετανάστευση και είναι σημαντικό να δοθεί επαρκή προσοχή σε αυτά για συμμετοχή τρίτων χωρών. Ερώτηση. Γιατί αποφάσισε να περιλάβει τρίτες χώρες σε αυτό το εσωτερικό χρηματοδοτικό μηχανισμό αντί να χρηματοδοτεί τις σχετικές δράσεις με εξωτερικούς ε, χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Και τώρα η διασύνδεση μεταξύ Κοινωνικού Ταμείου και AMF. Θέλετε να οριοθετήσετε τις αρμοδιότητες. Είδα όμως πριν ότι προβλέπονται εκπαιδεύσει γλωσσών. Αυτά μπορούν να χρηματοδοτούνται και από το Κοινωνικό Ταμείο. Από πού και μετά αρχίζει να χρηματοδοτεί το Ταμείο μετανάστευση και Ασύλου. Αυτά θα πούμε και αργότερα βέβαια. Τώρα σύντομα για τον μηχανισμό για τη χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό τελωνίων και συνοριοφυλακής. Οι εγκληματίες δεν έχουν βεβαίως κανένα πρόβλημα να βρουν που είναι ο πιο αδύνατος κρίκος των τελωνιακών ελέγχων. Σημαντικό η πρόταση λοιπόν, θα πρέπει να δούμε εάν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που χρησιμοποιεί η πρόταση είναι αρκετά καλά καθορισμένα και αντικειμενικά. Νομίζω εκεί μπορούν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις και να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην στήριξη που προσφέρουμε στις χώρες μέλη και σε ένα εναρμονισμένο τελωνιακό σύστημα στην Ένωση. Να διασφαλίσουμε επίση όμω ότι και οι χώρε μέλη εμπλέκονται επαρκώ στην ανάλυση και λήψη αποφάσεων σχετικά με, τα ποια μέσα, με το ποια μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε, ποια, σε ποιες διαβάσεις συνόρων. Ανάλυση κινδύνου, όγκων που διέρχονται τα σύνορα, όγκων εμπορευμάτων δηλαδή που διέρχονται τα σύνορα, να είμαστε βέβαιοι ότι ο μηχανισμός θα είναι αναλογικός και θα επιτρέπει αρκετή ευκαμψία ώστε να επιτυγχάνονται οι διάφοροι στόχοι. Αρκούμε σε αυτά και ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ. Έχουμε χρονικό περιορισμό, έχουμε και τον Επιτρόπο Κίνγκ, αλλά μιλούμε για άσυλο και μετανάστευση. Πώς είναι δυνατόν να υποτιμήσουμε την σημασία του θέματος, διότι είναι το μέγα θέμα σε αυτήν εδώ την κοινοβουλευτική θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βεβαίω νομικά αλλά και κυρίως πολιτικά. Αυτό είναι το μέγα θέμα, ξαναλέω. Θα εκτιμήσω πολύ την παρουσίασή σας, βεβαίως τεχνικές λεπτομέρειες, ωραίος ομορφότυπος που θα χρησιμοποιήσετε, αλλά ο ελίπων κρίκο είναι αυτός ο ελέφαντα μέσα στην αίθουσα. Δηλαδή, αλληλεγγύη. Και ναι, λέμε ωραία λόγια, ότι δήθεν το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης θα στηρίξει την αλληλεγγύη, όμως ε, το άρθρο 80 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλεί για αλληλεγγύη. Δεν είναι επομένω ευχολόγιο. Είναι ε, νομική επιταγή. Εμείς δεν βλέπουμε καμία διασύνδεση του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης με οποιαδήποτε αλληλεγγύη. Βλέπουμε να ε, είναι απελπισμένες οι χώρε πρώτης υποδοχής, οι οποίε ξαφνικά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή με τα λιμάνια υποδοχής σε οποιαδήποτε κρίση και πάντοτε συμβαίνει κάποιο επεισόδιο το οποίο αναμένεται να ακολουθήσει μετά από το προηγούμενο, τώρα είναι η Ισπανία. Πρώτο λιμάνι υποδοχής. Χρειαζόμαστε την αλληλεγγύη. Πού βρίσκεται η αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε. Πού βρίσκεται η ιδέα μιας ευρωπαϊκής κλίμακας αντίδρασης, όχι μόνο της χώρας που έχει βρεθεί σε απελπιστική κατάσταση. Πρώτα ήταν η Ιταλία. Έλλειψη αλληλεγγύης σημειώθηκε και εκεί και αυτός ο παράγοντας οδήγησε στην απόγνωση στην οποία βρίσκεται τώρα πλέον η Ισπανία. Καμία αλληλεγγύη λοιπόν, αλλά βέβαια κάπου γίνεται κάποια επίσημη παραπομπή ε, στην αλληλεγγύη, ίσως την πρώτη σας διαφάνεια, δεν ξέρω πού αλλού. Και το δεύτερο, πολύ σύντομα, βέβαια, μια παραπομπή που περιλήφθηκε άλλωστε και σε μια διαφάνεια που είδα πριν, για την πρόθεση της ενόμιμης μετανάστευσης. Η διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης. Τι σημαίνει αυτό. Ενώ μιλούμε για έλεγχο συνόρων, για έλεγχο προξενικών θεωρήσεων, για ηλεκτρονική τεχνολογία επικοινωνιών, για την αποτροπή της παρανομής μετανάστευσης, για την ενίσχυση των επιστροφών, είτε εθελοντικών είτε εξαναγκαστικών. Αλλά μιλούμε για εθελοντικές επιστροφές όταν κανείς έχει, κάποιοι από αυτούς έχουν διακινδυνεύσει τη ζωή τους για να φτάσουν ως παράτυποι μετανάστες δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούν εθελοντικά να επιστρέψουν. Δεν είναι επιλογή. Πάντοτε οι επιστροφές είναι αναγκαστικές. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αναγκαστικές επιστροφές. Αλλά δεν υπάρχει πάλι καμία διασύνδεση με κανένα παράθυρο ευκαιρίας για οποιαδήποτε νόμιμη οδό ώστε να μπορούν να έρχονται κάποιοι νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εξακολουθεί να υπάρχει αντίφαση. Διευρύνουμε διαρκώς το χάσμα ανάμεσα στις προσπάθειές μας. Να οδηγήσουμε σε αναγκαστικές επιστροφές τους παράδειγους μετανάστες, αλλά εγκαταλείπουμε την προσπάθεια να ανοίξουμε ένα νόμιμο δρόμο ώστε να φτάνουν κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, Επειδή δεν έχουμε χρόνο, συνάδελφοι, ε, και πρέπει να συζητήσουμε με τον Επίτροπο Κίνγκ, πρέπει να σχεδιάσουμε μια δεύτερη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό στην ΛΥΜΠΕ στις επόμενες εβδομάδες. Λυπούμε γι' αυτό, αλλά να ζητήσω τώρα από την Κομισιόν να μας δώσει μια απάντηση 10 δευτερόλεπτα. Τα, και τη συνέχεια γραπτός. Ναι, 10, λεπτά, 10 δευτερόλεπτα Βεβαίως για την αλληλεγγύη είναι ε, πάντα ευπρόσδεκτη, είναι παντού, σε κάθε κομμάτι αυτού του εγγράφου. Έχουμε στη ε, σελίδες 7, 16, 18, 21, 29 αναφορές ε, στην αλληλεγγύη. Έχει εξαφανιστεί ως στόχος, ναι, ως ρητό στόχος, διότι έχει ενταχθεί στους γενικούς στόχους. Έχουμε επανεγκαταστάσεις, μετεγκαταστάσεις, δράσεις, όταν θέλουν οι άνθρωποι να έρθουν εδώ στην Ένωση, ναι, στήριξη των κρατών μελών αλλά και των φορέων. Θα απαντήσουμε λοιπόν γραπτός. Οι ερωτήσεις ήταν εξαιρετικές όσον αφορά τους δείκτες, τα ποσοστά κτλ. κτλ. Λοιπόν, θα, δούμε, θα προσβλέπουμε στην επόμενη ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ και εγώ. Συνάδελφοι, να καλωσορίσω τον Επίτροπο Κίνγκ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα συζητήσουμε τις προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου. Η συζήτηση θα διαρθρωθεί Ε, καταρχάς θα έχουμε, ως εξής θα, έχουμε θα ακούσουμε πρώτα τον Επίτροπο και μετά θα έχουμε ερωταπαντήσει από εσάς. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Πριν από ένα χρόνο με καλέσατε για να σας αναφέρω ότι έχουμε κάνει για μια πραγματική και αποδοτική ασφάλεια στην Ένωση, στην πρώτη μου χρονιά ω Επίτροπο και αυτή ελπίζω να ήταν μια ε, χρήσιμη ε, ε, ανταλλαγή απόψεων. Ναι, βεβαίως ε, πρέπει να αντιμετωπίζουμε και να συλλαμβάνουμε τις απειλές. Ε, σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω, για, βέβαια για οποιοδήποτε θέμα θελήσετε, αλλά όλος ιδιαίτερος θέλω να αναφέρω τη διπλή της διπλή πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, δηλαδή να αποδώσουμε στις εξαιρετικές προτάσεις και να εφαρμόσουμε ε, αποτελεσματικά τα όσα ήδη έχουν ε, συμφωνηθεί. Γιατί αναγνωρίζουμε ότι υπήρχε μια διπεδηρίωδος όπου η Κομισιόν, ε, το Κοινοβούλιο και τα κάτι μέλη θα πρέπει πλέον να αποδώσουν, να δώσουν αποτελέσματα σε σχέση με τα όσα συμφωνήσαμε από κοινού να κάνουμε. Αναγνωρίζω ότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα στους επόμενους μήνες. Επίσης αναγνωρίζω ότι υπάρχουν ίσως κάποια κενά ή φραγμοί στους τομείς πολιτικής, ας πούμε όπως τονίζεται στην, στην έκθεση πώς ε, το κόστος της μη ύπαρξης Ευρώπης στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ας κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω όμως για να θυμίσουμε ότι πώς μάλλον οργανώσαμε την εργασία μας σε αυτό το τομέα για να, να, να αντιμετωπίσουμε την απειλή της τρομοκρατίας έχουμε κάνει μια διπλή προσέγγιση. Καταρχάς να κλείσουμε τον χώρο που χρειάζονται όσοι θέλουν να μας βλάψουν και φτιάχνοντας αντοχή ανθεκτικότητα απέναντι σε επιθέσεις. Ε, συνεργαζόμαστε ώστε να κλείσουμε το χώρο που χρησιμοποιούν οι τρομοκρατές ε, περιορίζοντας το ε, δυνατότητά τους να κινηθούν, να έχουν χρήματα, να βρουν εξοπλισμούς πυρομαχικά αλλά και εργατικό δυναμικό. Έχουμε κάνει αυστηρούς ελέγχους στα σύνολα για να μπορέσουμε να συλλάβουμε αυτούς που χρησιμοποιούν ψεύτικες ταυτότητες. Όπως είπαμε τα δεδομένα είναι θέμα κλειδί σε, αυτή μας, σε αυτό μας τον αγώνα. Εργαζόμαστε ώστε να βελτιώσουμε τα συστήματα που υπάρχουν, να είναι διαλειτουργικά και να μπορέσουμε να καλύψουμε και κάποια κενά ενημέρωσης και πληροφοριών. Γι' αυτό έχουμε το React, το ETIA, το EQUES, έχουμε ενημερώσει το SIS και ούτω καθεξής για να μην μπορούν οι τρομοκράτες να έχουν πρόσβαση στα χρήματα που χρειάζονται, έχουμε κάνει την τέταρτη και πέμπτη οδηγία κατά του ξεπλήματος χρήματος και ε, όσον αφορά τα όπλα και το πυρομαχικά έχουμε ενισχύσει του ελέγχου για τα ε, πυροβόλα όπλα, εισαγωγές και εξαγωγές, αλλά και ε, να περιορίσουμε ε, τα κρυκτικά για να εμποδίσουμε τον ΤΑΕΣ και τους άλλους να έχουν το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται. Λάβαμε μια σειρά από μέτρα για να ενισχύσουμε την εργασία μας και μάλλον ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την εργασία μας για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Δεύτερος ε, κλάδος, δηλαδή η οικοδόμηση ανθεκτικότητας, θέλουμε να προστατεύσουμε καλύτερα τους δημόσιους χώρους μας, και έχουμε διαθέσει και πόρους ε, εκτός από τη συνεργασία. Θέλουμε, έχουμε βελτιώσει την ασφάλεια στους σιδηροδρόμους αλλά και όσον αφορά τον κίνδυνο χημικής και βιολογικής ε, ε, ε, επιθέσεως που δυστυχώς κατέστη προφανής μέσω των επιθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο νωρίτερα φέτος. Ο πρόεδρος Γίνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωση είπε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις κυβερνοαπειλές και έχουμε κάνει πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία της, του οργανισμού για την, ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για ε, την κυβερνοπροστασία να εξασφαλίσουμε και τις διαδικασίες τις εκλογικές μας Ποια είναι λοιπόν τα θέματα κλειδιά που τώρα βρίσκονται επιτάπητες, ποιες είναι οι νομοθετικές προτάσεις ε, που από κοινού θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Πρώτον, οι προτάσεις μας να καταστήσουμε τα, προγράμματα, τα, τα συστήματα πληροφοριών διαλειτουργικά. Ε, είναι, ο κύριο Λέναρτς είναι ο εισηγητή. Έχουμε χίλιε τροπολογίες που κατατέθηκαν από τα μέλη. Ξέρω πω οι εισηγητέ εργάζονται σκληρά για να προετοιμάσουν συμβιβαστικέ. Εγώ και η ομάδα μου είμαστε έτοιμοι να σα στηρίξουμε στο να προχωρήσει αυτή η δουλειά ε, όσο γίνεται καλύτερα. Ε, ο κύριος Λέναρ και ο κύριος Μέλο είναι οι ε, ε, και προσβλέπουμε στην γρήγορη ε, διεκπαιρέωση αυτής της έκθεσης. Έπειτα, αστυνομικές και δικαστικές αρχές να έχουν και μαρτυρίε, ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία με σερβασμό στα θεμελιώδη ανθρωπίνα δικαιώματα. Και μάλιστα οι προτάσει αυτέ είναι βελτίωση, όπου τα εθελοντικά κανάλια συνεργασία μπορεί να είναι ελληματικά όσον αφορά τη διαφάνεια και την ε, διαλειτουργικότητα. Θέλουμε να βοηθήσουμε και εδώ έχουμε την κυρία Σίπελ ως ε, εισηγήτρια και ελπίζω πως τα σχετικά μέτρα θα υιοθετηθούν πριν το τέλος τη τρέχουσα θετίας. Πρότασή μας για ενίσχυση των ισχυών των κανόνων για την ε, διαφήμιση και τη χρήση εκρηκτικ... εκρηκτικών και εδώ ελπίζουμε να υπάρξει συμφωνία πριν το τέλος αυτής της θητείας. Τέταρτον, πρόταση να καταστήσουμε δυσκολότερη την μεταφορά ε, κονδυλίων για, ανάμεσα σε λογαριασμούς και κράτη για τους τρομοκράτες, δίνοντας ε, πρόσβαση στη, στα Μητρώα των κεντρικών τραπαζών. Ε, ελπίζουμε πως αυτές οι προτάσεις θα εξεταστούν σύντομα ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα εδώ στις συζητήσεις στο Κοινοβούλιο. Επομένως, ε, στην ε, συνεργασία με τον εισηγητή Ράντοφ. Ε, δυνατότητα αντιμετώπιση απατών που δεν αφορούν μετρητά από τι αστυνομικέ αρχέ των κρατών μελών. Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με το Κοινοβούλιο, ώστε η τελική εκδοχή τη οδηγία να ενισχύσει τη δυνατότητα αντιμετώπιση αυτών των εγκλημάτων. Ε, των αδικημάτων. Ε, μετά, εισηγητής κυρία Δεπρέ ε, θέλει να αντιμετωπίσουμε τη χρήση των πλαστών εγγράφων που χρησιμοποιούν τρομοκράτες και εγκληματίες. Τώρα, κυβερνοαπειλές που θα σας απασχολήσουν επίσης και θα ήθελα να θυμίσω ότι η Κομισιόν εργάζεται τώρα σε μια για μια πρόταση για την αντιμετώπιση, νομική αντιμετώπιση τρομοκρατικού ε, περιεχομένου online. Ε, έχουμε αντιμετωπίσει με το EU Internet Forum τους τρομοκράτες ε, στο ίντερνετ και καταφέραμε αρκετά μέσω της εθελοντικής συνεργασίας, αλλά ακόμα πρέπει πολλά να γίνουν, γιατί υπάρχει ακόμα πολύ τέτοιο περιεχόμενο στο ίντερνετ. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την, ε, την και να δώσουμε μάλλον περισσότερο feedback για να μπορέσουμε να φτιάξουμε σχετική νομοθεσία όπως ζήτησε ε, το Συμβούλιο αλλά και το Κοινοβούλιο για τις ε, πλατφόρμες τις Ιντερνετικές και την ψηφιακή αγορά. Ως αποτέλεσμα αυτών των αυτών όλων θα σας ε, έρθουν διάφορες νομοθετικές προτάσεις. Τέλος, για τη συνεργασία που έχουμε συζητήσει και παλιότερα, η ανάγκη να συνεχίσουμε αποτελεσματικά για τα όσα συλλογικά συμφωνήσαμε να κάνουμε. PNR. Ε, συζητήσαμε το PNR επανειλημμένα η προθεσμία για μεταγραφή της οδηγίας ε, ε, εξέπνευσε το Μάιο. Εμείς ε, τον Ιούλιο ξεκινήσαμε διαδικασίες κατά παράβαση ενάντια στις χώρες που δεν είχαν πλήρως εφαρμόσει την οδηγία. Τώρα έχουμε 17 κρατη που έχουν κοινοποιήσει την πλήρη μεταγραφή. Δύο ακόμα έχουν κοινοποιήσει την μερική και αναμένουμε και άλλοι να κοινοποιήσουν προσεχώς. Τώρα χρειάζεται να κάνουμε νέες δράσεις για την εφαρμογή της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων ε, από την αστυνομία και εδώ ξεκινήσαμε διαδικασίες κατά παράβαση τον Ιούλιο ασφάλεια είναι η πρώτη μας νομοθεσία γιατί θα βελτιωθούν οι δυνατότητες σε εθνικό επίπεδο, θα αυξηθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία και θα εξασφαλιστεί η διαχείριση του κινδύνου καθώς και οι δυνατότητες ε, ε, αναφορών ε, για όλους τους φορείς ψηφιακών υπηρεσιών και η οδηγία για τη συνεργασία που αφορά την αστυνομική συνεργασία για την προστασία των δεδομένων για την πρόληψη, έρευνα και δίωξη των εγκλημάτων. Έτσι, οι αστυνομικέ αρχέ θα κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά του, ενώ θα προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτά είναι κλειδιά ε, για την ε, κοινή μας ασφάλεια. Πρόκειται για μέτρα τα οποία έχουν ε, κοντινές ε, προθεσμίες, 8 Σεπτεμβρίου για η οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η οδηγία για τα πυροβόλα όπλα στις, 15 ε, Σεπτεμβρίου. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να εξασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή αυτών των οδηγιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτού του είδους απειλές ε, όταν αρχικά σας ε, είδα ως ε, ένας ταπεινός υποψήφιος επίτροπος ε, και σας είχα πει ότι οι τρομοκράτες αλλά και έγκλημα βασίζονται στην έλλειψη του συντονισμού μεταξύ των κρατών. Από ό,τι φαίνεται δεν θα με δώσει ένα χρόνο για να σας πω ποια πρόοδος έχει σημειωθεί, αλλά σε διάρκεια των επόμενων 7 μηνών θα είμαι πεπισμένος και είμαι ε, προσιλωμένος στο να μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε ε, ό,τι μπορούμε περισσότερο σε όλα τα μέτωπα που έχουμε θέσει μπροστά μας για, ως στόχους για να εξασφαλίσουμε ασφαλή Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους μας τους πολίτες. Πρόεδρος. Αρχίζει το γύρο των ερωτήσεων. Δύο λεπτά. η κυρία Μετσόλα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ και μας κάνατε την παρουσίαση. Δεν θα χρειαστώ δύο λεπτά. Θα ήθελα να μας δώσετε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάχρηση των προσωπικών δικτύων από τα κοινωνικά δίκτυα και αυτό πριν από τις ευρωεκλογές. Αναφέρομαι ιδιαίτερα σε αυτά τα οποία είχατε πει το καλοκαίρι ότι κάποιες διαδικασίες που παρεμποδίζουν τις δημοκρατικές διαδικασίες είναι βασική μας ανησυχία στο μέλλον. Αυτό απαιτεί άμεση δράση και συνδέεται με τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εκλογείς μας. Τι θα κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ. κυρία Σίπελ. Ένα τομέα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, που έχει ήδη τεθεί βέβαια. Οι αστυνομικές αρχές επίσης αλλάζουν. Αλλάζουν και προσπαθούν να καλύψουν τις νέες εκφάνσεις της εγκληματικής δραστηριότητας. Είναι σαφές ότι και μετά από τις πρώτες εξτρεμιστικές επιθέσεις συγκεντρώσαμε την προσοχή μας στην καταπολέμηση των τρομοκρατικών ενεργειών. Ταυτόχρονα υπήρξαν και κάποιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι τρομοκράτες, στον τρόπο με τον οποίο την χάνουν στήριξης οικονομικής, ε, στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η ριζοσπαστικοποίηση των κρατουμένων είναι σαφές λοιπόν ότι απαιτούνται συμπληρωματικά μέτρα. Ε, διαρωτώ με αν θα μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι και προσαρμοστικοί σε τέτοιες αλλαγές. Τα τελευταία χρόνια οι επιθέσεις ε, από πλευράς των, Ισλαμικών, των Ισλαμιστών τρομοκρατών αλλά είδαμε αύξηση όμως ακραίων ενεργειών από ακροδεξιές και ακροαριστερές ομάδες. Αυτού του τύπου λοιπόν οι διαφορετικές επιθέσεις που είναι διαφορετικής προέλευσης μήπως χρειάζονται διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης σε σχέση με τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα για τα κοινωνικά μέσα και τις ευθύνες που έχουν. Εδώ έχω αρκετές ανησυχίες. Μιλάμε για παγκόσμιους εταίρους που παρουσιάζουν ή αποκρύβουν σε παγκόσμια κλίμακα τα γεγονότα. Εμείς κατά κάποιο τρόπο έχουμε επιτρέψει να ιδιωτικοποιηθεί η λήψη αποφάσεων γύρω από το τι θα συμπεριλαμβάνεται και τι θα αποκλείεται από τον ψηφιακό κόσμο υπάρχει απάντηση στον τομέα αυτό. Βλέπουμε πάρα πολύ συχνά ότι αυτό το οποίο διαγράφεται από το διαδίκτυο ε, δεν γίνεται με τον σωστό τρόπο και ε, δεν γίνεται και από αλγορίθμους μόνο. Γίνεται από εκατοντάδες και χιλιάδες υπαλλήλους κάτω από συνθήκες εργασίας απαράδεκτες το θέμα είναι λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε με τις επιχειρήσεις αυτές, πώς μπορούμε να διακανονίσουμε τον τρόπο λειτουργίας τους και πώς, και αυτή είναι μια γενική ερώτηση, όχι μόνο προς την Επιτροπή, να μπορέσουμε να ελαχιστοποιήσουμε την δύναμη και την εξουσία των μεγάλων αυτών επιχειρήσεων ε, έτσι ώστε να μην είναι ε, ιδιωτική απόφαση το ποια μηνύματα είναι αυτά τα οποία θα αποστέλλονται και ποια όχι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τερικάμπρας. Έχω τρεις ερωτήσεις επίτροπε. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε σχετικά συνοπτικά το τι θα περιλαμβάνει ο επόμενος κανονισμός για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου online που θα δημοσιεύσετε στις 12 Σεπτεμβρίου επισήμως. Δεύτερον, πώς θα διασφαλίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η έβρεση περιεχομένου το οποίο είναι παράνομο δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με το περιεχόμενο το οποίο απαρέσκει σε ορισμένους. Ποια είναι η διαφορά και τα σύνορα ανάμεσα στην προστασία από τη μία και τη λογοκρισία από την άλλη. Από την άλλη, πώς μπορούμε αυτοί οι οποίοι φορτώνουν τέτοιου είδους περιεχόμενο θα μπορούν να διώκονται πώς μπορούμε να, πώς μπορούμε να τους παραπέμψουμε όταν οι αποδείξεις των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων διαγράφονται. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ που συνοψίσατε το έργο σας των τελευταίων ετών αφής ε, αναλάβατε. Είναι σημαντικό πράγματι για να εξασφαλιστεί και εφαρμογή από τις χώρες μέλη. Σας ερωτώ τώρα. Συζητούμε έκθεση για την τρομοκρατία. Σας ερωτώ λοιπόν. Ποια είναι η γνώμη σας για τις διάφορες προτάσεις του σχέδιου εκθέσεως για τη δημιουργία νέων θεσμικών οργάνων, νέων οργανισμών δεν υπάρχει κίνδυνος ε, επικάλυψης. Για παράδειγμα, εδώ για το κέντρο υπεροχής κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Μήπως μπορεί απλώς να σημαίνει μια αναβάθμιση του ραν τώρα για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Γνωρίζω ότι οι χώρες μέλη δεν έχουν τηρήσει ακόμη τα υπεσχημένα σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ. Επιτρέπουν ακόμη δηλαδή και σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατικές και το ύψος των δράσεων αυτών υποστηρίζεται από τον Μοσκοβισή στα 50 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πραγματικά ε, ε, τρομερό. Θα ήθελα να το δείτε αυτό υπό την οπτική γωνία της ασφάλειας. Και σα ρωτώ επίσης κάτι που αναφύεται όλο και, αναδύεται μάλλον όλο και πιο ανάγλυφα, ότι δηλαδή μαφίες εμπλέκονται στην διακίνηση ανθρώπινων όντων και βέβαια και τρομοκρατικές οργανώσεις και ε, η χρηματοδότηση εκεί παίζει ένα σημαντικό ρόλο και οι χώρες την διώκουν. Και τέλος ε, ο ρόλος των κρυπτονομισμάτων. Πώς βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο τα κρυπτονομίσματα εμφανίζουν τώρα ε, μια εικόνα πιο μεγαλύτερης έγκλης. Ε, κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ελέγξει την ε, εξέλιξη αυτή. Και επίσης μη επανδρομένα αεροσκάφη, αυτόνομα οπλικά συστήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Ήδη τα επανδρομένα αεροσκάφη μπορεί να μας παρακολουθούν και μάλιστα χρησιμοποιούνται και σε εγκληματικές δραστηριότητες. Θα προχωρήσουν σε ένα επόμενο στάδιο τεχνητής νοημοσύνης η οποία θα χειρίζεται τα αυτόματα οπλικά συστήματα. Σας ερωτώ τέλος. Μπορείτε να μας πείτε ποιες χώρες μέλη ανθίστανται στην ε, διαδικασία επί παραβιάση για την οποία αναφερόμαστε. Κύριος Ντεπρέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πρώτα τον Επίτροπο. Που είναι πάντοτε στη διάθεσή μας όταν το, το ζητούμε. Ενδιαφέρουσα άλλωστε εμπειρία που για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει χαρτοφυλάκιο επιτρόπου ειδικό για την ασφάλεια. Και έχει κάνει και η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την σύσταση να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον. Εξηγήσατε τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί. Έχω τώρα κάποια σχόλια. Πρώτο, διαλειτουργικότητα Νομίζω ότι θα πολλαπλάσιαζουμε τις προσπάθειες για να φτάσουμε σε κάποια συνένεση, γιατί είναι από τα βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής των πληροφοριακών συστημάτων που έχουν δημιουργηθεί και χρειάζεται πολλαπλασιασμός των προσπαθειών, όπως είπα. Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία ασφαλείας στις ε, ταυτότητες, στα δελτία ταυτότητας. Έχουμε τις ε, σχετικές εκθέσεις από FRA και EDPS και νομίζω ότι στη βάση αυτή μπορούμε να προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση. Έχω τώρα ερωτήσεις για τα ζητήματα που αναφέρατε. Πρώτα, σχετικά με το τρομοκρατικό περιεχόμενο επιγραμμικά, στο διαδίκτυο δηλαδή. Πότε θα περάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απειλή λήψη μέτρων. Εγώ λέω, παρά τις δυσχέρειες, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν δυσχέρειες, και τεχνικές και νομικές και σεβασμού δικαιωμάτων. Τι σας έκανε να αλλάξετε άποψη ωστόσο. Τέλος, η κρυπτογράφηση. Εγώ διαβάζω διάφορες πληροφορίε και βλέπω ότι στο επίπεδο της Κομισιόν διεξάγονται συζητήσεις και κατατίθεται προτάσεις για, μια, για ένα οργανισμό όπως η Ευρωπόλ. Τι γίνεται με την κρυπτογράφηση. Και ένα θέμα πολυτεχνικό. Για τις διευθύνσεις IP, διότι η, η υπηρεσία ασφαλείας περνούν ατέλειωτο χρόνο για να διαπιστώσουν ποιες ε, διευθύνσεις είναι ύποπτες. Ενώ υπάρχει τρόπος, υπάρχουν συστήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτεχνηθεί η διαδικασία αυτή. Και τέλος, προετών, όταν συζητούσαμε για την εισαγωγή ενός συστήματος όπου είχε προσκρούσει σε πολλές ε, επικρίσεις. Από τότε που ισχύει ωστόσο το IPR στην χώρα μου, 13 άτομα διώχθηκαν στην βάση του, ε, της χρήσης του συστήματος PNR, δηλαδή της ε, δήλωσης των προσωπικών στοιχείων των επιβατών αεροπορικών εταιριών. Παρατήρηση χωρίς μικρόφωνο. Αυτά είχα να πω κύριε Επίτροπε. Βεβαίω οφείλω να διατηρώ και εγώ την αίσθηση του χιούμορ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κάτι είπε ήδη η κυρία Ζίπελ προηγουμένως για την τρομοκρατία του Ισλάμ. Από την άλλη μεριά αυτό που βλέπουμε είναι άνοδος της βίας της άκρας δεξιάς, κηρύγματα μίσους, επιθέσεις κατά μεταναστών ή ε, κατά προσφύγων. Είδαμε και στη Γερμανία τι έγινε τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η ε, άνοδος της βίας της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη. Δεύτερο, διαλειτουργικότητα. Ω και ο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Ούτε βέβαια πρόκειται να κάνω εδώ σαν να είναι συνάντηση σκιωδών εισηγητών για το θέμα αυτό, αλλά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το τι σημαίνει διαλειτουργικότητα. Σύμφωνα με τη δική μα κατανόηση, η διαλειτουργικότητα σημαίνει να επιτρέπουν να επιτρέπεται, να διευκολύνεται η επικοινωνία μεταξύ των υφισταμένων τραπεζών δεδομένων. Αυτό είναι σημαντικό θέμα. Θα το συζητήσουμε με τους μου και την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, γιατί κατά τη γνώμη μας δεν χρειαζόμαστε αυτό το Common Identity Repository. Έχουμε το BMS, έχουμε άλλους φορείς, άλλα, ε, άλλους και τράπεζες δεδομένων που νομίζω δεν χρειάζεται τελικώς το Common Identity Repository. Αυτό το συζητήσουμε και στους κοιοδησίγητες, αλλά σας ρωτώ, σας παρακαλώ να μας εξηγήσετε πώς βλέπετε τις διαφορές αυτές για το Common Identity Repository. Η ε, κυρία Τσίνιτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τον Επίτροπο Κιν για την παρουσία του εδώ και τις προσπάθειες τις οποίες κάνει στον τομέα της ασφάλειας και τις οποίες γνωρίζουμε καλά και με τις οποίες φυσικά συμφωνούμε και στηρίζουμε. Πολλά από αυτά που ήθελα να πω καλύφθηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές και με την παρατήρηση κυρίως της κυρίας Γκομές για τα θέματα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τη σχέση τους με τη μαφία και το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει αντιμετωπιστεί νομίζω πολύ προσεκτικά και δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη αυτή πλευρά των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Τώρα για το θέμα της ριζοσπαστικοποίησης και της πρόληψης της. Θα ήθελα την άποψή σας γι' αυτό γιατί είναι ένα κεντρικό θέμα και τίθεται το θέμα επίσης των παρεμβάσεων σε επίπεδο ε, των συστημάτων εκπαίδευσης για την αποτροπή του συγκεκριμένου φαινομένου. Και υπάρχουν επίσης και κάποιες ερωτήσεις λίγο πιο συγκεκριμένες σχετικά με την ομοθετική πρόταση η οποία προβλέπει ε, τα μέτρα που θα ληφθούν σε σχέση με το περιεχόμενο ε, των, ε, ε, των στοιχείων τα οποία φορτίζονται στο ίντερνετ. Είπατε ότι έχουν υπάρξει αποτελέσματα αλλά πολλά μένει ακόμα να γίνουν. Υπό το φως αυτής της παρατήρησης θα ήθελα να μου πείτε εάν πιστεύετε ότι η παρούσα πρόταση θα μπορούσε να προσφέρει κάτι έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. τι εγγυήσει μπορούμε να έχουμε ε, στα πλαίσια της πρότασης αυτής ε, για να φροντίσουμε από τη μία την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και να διασφαλίσουμε από την άλλη την ασφάλεια των χρηστών αυτά τα οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα στο ίντερνετ δεν ήσαν ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τον κίνδυνο το περιεχόμενο το οποίο διαγράφεται από μία πλατφόρμα να αναπαράγεται σε μία άλλη. Και υπό το φως της πρότασης αυτής διαρωτώ με ποιος θα είναι ο ρόλος της μονάδας στην οποία έχουμε και η οποία μέχρι τώρα λειτουργεί με χρήσιμο τρόπο για τον εντοπισμό της, των επικίνδυνων ιστοσελίδων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την παρουσία του, για τη διαλειτουργικότητα τώρα. Θα συνεχίσω το σκεπτικό του Επιτρόπου για την πρόταση αυτή, είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικά δεν ξέρω τι διαφορές απόψεως, απόψεων υπάρχουν και αν είναι τόσο ε, βαθιές όπως φάνηκε σε ορισμένες περιπτώσεις αλλά τους επόμενους μήνες θα τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά και ευχαριστώ και για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών σας που μας βοηθούν ιδιαίτερα σε σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων αυτών των θεμάτων τα οποία θέσατε. Τώρα για τα PNR, ε, μιλήσατε και για τις προσφυγές επί παραλήψη. Η οδηγία για το PNR είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο και είχε ληφθεί ε, άτυπη απόφαση από το Συμβούλιο ότι θα αντιλαμβάναμε υπόψη. Συνεπώς λοιπόν υπάρχουν κάποιες φήμες ότι ορισμένες χώρες έχουν αμφιβολίες για τη συμπερίληψη και των ενδοκινοτικών πτήσεων στις διαδικασίες του PNR. Θα θέλα λοιπόν τις απόψεις σας σχετικά με την λειτουργία του συστήματος αυτού στο σύνολό του και όχι μόνο για το θέμα το οποίο έχει ήδη συζητηθεί στο Συμβούλιο για τις ενδοκινοτικές πτήσεις. Τώρα πιστεύω ότι η Ιεροπόλη θα παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ως προς αυτό. Εξεπλάγει ακούγοντας ότι ο προϋπολογισμός για το 19 που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μειώνει κατά 21 εκατομμύρια ευρώ και 30 θέσεις από το οργανόγραμμα σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν αποφασίσει τα κράτη-μέλη στα πλαίσια της Διαχειριστικής Επιτροπής της Ευρωπόλης. Αυτό είναι ένα πολύ ανησυχητικό μήνυμα σε σχέση με τις προτεραιότητες τις οποίες χρειάζεται να αναλάβει η Europol. Ο Λόπες Θα ήθελα να συμφωνήσω και με τα υπόλοιπα μέλη τα οποία εξέφρασαν τις ανησυχίες τους γύρω από την σημαντικότατη κατά τα άλλα πρόταση που κάνετε για την ταχεία διαγραφή και αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Απαιτείται ένα νομικό πλαίσιο και απαιτείται ένα νομικό πλαίσιο έτσι ώστε ε, να ληφθούν οι απαιτούμενες κυρώσεις. Έχουμε και τη νέα αντιτρομοκρατική οδηγία αλλά απαιτούνται ε, νομικές αλλαγές και εξελίξεις ε, σε επίπεδο εθνικών νομοθεσιών Μερικές φορές όχι μόνο υπάρχουν διαφορετικού τύπου απαντήσεις, αλλά υπάρχει και πλήρης έλλειψη απαντήσεων σε σχέση με τον τρόπο αφαίρεσης του περιεχομένου. Και πολλές φορές υπάρχει και το θέμα της έλλειψης επιθυμίας συνεργασίας από πλευράς των παρόχων. Θα ήθελα λοιπόν τα σχόλιά σας για τις ιδέες τις οποίες έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το κομμάτι της προβληματικής και επιτέλους οι προτάσεις μας να καταστούν δράσεις. Σας ευχαριστώ λοιπόν για όλες τις ερωτήσεις σας. Θα ήθελα με ευχαρίστηση τώρα να δώσω το λόγο πάλι πίσω στον Επίτροπο. Ευχαριστώ. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα μπορέσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις στον χρόνο που, μου, που έχω. Αν δεν προλάβω θα σας δώσω γραπτά τις απαντήσεις. Θα σας στείλω γραπτά τις απαντήσεις. Για κάποια ζητήματα που προέκυψαν επανελειμμένα ε, θα προσπαθήσω να τα ομαδοποιήσω και να τα απαντήσω πρώτα. Για το θέμα του κατά πόσο ανταποκρινόμαστε στην ε, μεταλλασσόμενη φύση των απειλών που δεχόμαστε. Πρώτα το έθιξε η κυρία Σίπελ και μετά και άλλοι. Ελπίζω πως ε, από κοινού θα τα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό. Η μετακίνηση στη φύση της απειλής, της Ισλαμικής ε, ακραίας απειλής είναι, όπως το είπε η κυρία Σίπελ, πρόσφατα αντιμετωπίσαμε μια σειρά από μοναχικές επιθέσεις ανθρώπων που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί ή αυτο ριζοσπαστικοποιηθεί που χρησιμοποίησαν πολύ απλά πράγματα ε, μέσα για να σκοτώσουν πολίτες της Ένωσης και πρέπει να προσαρμοστούμε στο πώς θα απαντήσουμε σε αυτό και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε μέσω της εστίασης στην ε, ριζοσπαστικοποίηση και την προτεραιότητα σε που δίδουμε στην αντιμετώπιση της online ε, ριζοσπαστικοποίηση, ε, εστιάζουμε σε αυτό γιατί είναι αποδεδειγμένο δυστυχώς ότι είναι αποτελεσματικό το, το, το περιεχόμενο ε, που υπάρχει online για να ριζοσπαστικοποιηθούν οι νέοι άνθρωποι. Τώρα βέβαια θα πρέπει να ξαναδούμε κατά πόσο έχουμε χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να το καταφέρουμε αυτό ή όχι. Ε, να το σκεφτούμε λοιπόν αυτήν την μεταβαλλόμενη απειλή και να δούμε κατά πόσο η εργασία μας για τη ριζοσπαστικοποίηση έχει εστιαστεί αποκλειστικά ε, σε αυτήν. Εγώ συμμετείχα σε συνεδριάσεις και συζητήσεις για το να έχουμε πιο αποτελεσματικά μέσα να αντιμετωπίσουμε και άλλες μορφές ριζοσπαστικοποίησης από οποιοδήποτε άκρο και από την άκρα δεξιά. Συνειδητοποιώ ότι αυτό του είδους ε, οι ακρότητες μπορεί να οδηγήσουν ε, σε, σε, σε δολοφονίες όπως η Τζο Κόξ που ήταν μέλος του Κοινοβουλίου ε, είναι ένα παράδειγμα. Έχουμε κάνει λοιπόν δουλειά με τους εμπειρογνώμονες ώστε να μπορέσουμε να ανανεώσουμε τις προσπάθειές μας κατά της ρωσπαστικοποίησης αλλά και με τον εξωτερικό έλεγχο που μας ασκείται το ελεκτικό συνέδριο επίσης έχει κάνει μια σχετική έκθεση και όλα αυτά είναι ευπρόσδεκτα προσπαθούμε να αλλάξουμε τη διοργάνωση τη δουλειά μας για την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης μέσα στην Κομισιόν και προσβλέπω σε νέες ευκαιρίες για να το συζητήσουμε πρόκειται για την Ισλαμική εξτρεμιστική απειλή ε, και άλλες τρομοκρατικές απειλές που υπάρχουν τώρα. Θα προτείνουμε κανονισμό. Φοβούμαι ότι θα πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή για τις λεπτομέρειες, γιατί η ανακοίνωση προβλέπεται για την επόμενη εβδομάδα. Ευχαρίστω θα επανέλθω για να συζητήσουμε αυτή, ε, την, συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση για τις λεπτομέρειες από τη στιγμή που θα έχουν κατατεθεί οι προτάσεις. Με τα χαρά θα το κάνω. Ελπίζω πως όταν θα δείτε τις προτάσεις θα έχετε υπόψη το πλαίσιο και θα έχετε επίσης ε, τη δυνατότητα να το δείτε επί τη βάση της προόδου που έχουμε κάνει ε, στην συνεργασία αλλά και τις προκλήσεις που έχουμε αντιμετωπίσει με τις πλατφόρμες που ακόμα δεν έχουμε λύσει. Δηλαδή, ξεκινήσαμε με μια προσέγγιση το περασμένο Σεπτέμβριο, με περισσότερες λεπτομέρειες στη σύσταση τον Μάρτιο και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να κλείσουμε όλα τα κενά και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που εντοπίσαμε και με τις ε, πλατφόρμες. Δεν έχουμε ακόμα δηλαδή αποτελεσματική βάση για να αντιμετωπίζουμε ε, περιεχόμενο μας αναφέρεται. Όταν λοιπόν η επιβολή του νόμου και αυτό απαντώ στην κυρία Κινίτσι για το ρόλο των IIU όχι μόνο στην Ένωση αλλά και στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να έχουν IIU. Δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη ακόμα μονάδες αναφορές. Δηλαδή, όταν οι αστυνομικές αρχές αναφέρουν ε, παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο, τότε θα πρέπει να δράσουμε και πρέπει να θεσπίσουμε μια βάση για να δράσουμε. Επίσης, πρέπει να θεσπίσουμε σαφή και διαφανείς νόμους για τη χρήση ε, αυτοματοποιημένων μέσων που χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους. Χρειάζονται σαφήνεια εδώ για να αντιμετωπίσουμε και τις ανησυχίες για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειάζεται συνεργασία, επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στις πλατφόρμες και ε, συνεργασία με τις, αρχές, ε, τις Αυτά λοιπόν θα θέλαμε να τα συζητήσουμε μαζί σας πιο λεπτομερώς, αν το επιθυμείτε κι εσείς. Ε, τώρα, πολύ ε, τώρα συμμετείχατε στην Επιτροπή και προσβλέπω να σας δώσω αυτό το πλαίσιο για να συζητήσουμε για τις προτάσεις και τις λεπτομέρειές τους για το, τη συγκεκριμένη ερώτηση της κυρίας Γκόμες για το κατά πόσο υπάρχει επικάλυψη. Ελπίζω πως όχι. Ας πούμε, για το πώς οργανώνουμε τη δουλειά μας για την ριζοσπαστικοποίηση, ναι, σίγουρα μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Να μάθουμε από αυτά που έχουμε κάνει και να βελτιώσουμε την οργάνωσή μας. Για αυτό το θέμα, όχι μόνο της ε, ολοκλήρωσης των κρεμών προτάσεων. Σας ευχαριστώ όλους όσους μιλήσατε για τη σημασία της προόδου στις εκκρεμείς αυτές προτάσεις, για τις ταυτότητες, τη λειτουργικότητα. Ε, επίσης δεν θέλω να ξεχνάμε την εφαρμογή. Ξέρω πως δεν θα με αφήσετε να το ξεχάσω. Κάνουμε τακτικές εκθέσεις. Κάνουμε ε, πολλές δραστηριότητες. Αν υπάρξει οποιοδήποτε θέμα, ε, ζητήστε μου και θα απαντήσω εννοείται. Ρωτήστε με και θα απαντήσω. Για τη Europol δεν θα πρέπει να αμφιβάλλετε. Ξέρετε ότι η συζήτηση για τον προπολογισμό συνεχίζεται. Απλώς επιστώνω το αντικειμενικό γεγονός ότι αυτό που συνήθως γίνεται είναι ότι ο προπολογισμό προχωρά και περνάει. Και αυτό αντικατοπτρίζει την σημασία που έχει η Europol μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το θέμα της διαλειτουργικότητας τέλος, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που, που, είχαν ε, αναφερθεί. Ε, προσβλέπω στη στενή συνεργασία και ε, βλέπω και συμφωνώ με τον κύριο Τεπρέ πως πρόκειται για βασικό λίθο στην αρχιτεκτονική που προσπαθούμε να κατασκευάσουμε από κοινού. Ε, είμαστε θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των συστημάτων που έχουμε. Ε, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση λοιπόν για τις λεπτομέρειες και για το κοινό αποθετήριο ταυτοτήτων. Είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο των προτάσεών μας. Δεν είναι όπως είπα συλλογή νέων δεδομένων, ούτε αποθήκευση νέων δεδομένων. Δεν δημιουργούνται νέοι κανόνες για την πρόσβαση στα δεδομένα, πρόκειται για αποτελεσματική αναζήτηση. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, αλλά και η συζήτηση και σε οποιοδήποτε σημείο για τις, από των εκκρεμών ε, προτάσεων, με στόχο να φτάσουμε σε συμφωνία μαζί σας μέσα σε αυτή την εντολή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κίνγκ, Επίτροπε Κίνγκ. Ευχαριστώ για την αφήξή σας εδώ και για τη συζήτηση για το νέο κανονισμό. Σε ευχαριστώ και για την πληρότητα των απαντήσεων. Okay, dear colleagues. Uh, Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ας προχωρήσουμε τώρα λοιπόν στο υπαριθμόν 9 της ημερησίας διατάξεως εξέταση του σχεδίου εκθέσεως των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το έτος 2017. Ο κ. Τερικάμπρας είναι εισηγητής. Πρόκειται για ή έκθεση, αντιπροσωπευτική του έργου της Επιτροπής μας, καλύπτει ευρύ, θέσμα θεμάτων, ευρύ φάσμα θεμάτων, προκλήσεις των, της, του σεβασμού των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων των προσώπων που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Τερικάμπρας, έχετε το λόγο. Πρώτα, ζητώ συγγνώμη, διότι Είμαι εδώ μαζί σας από τις 9 το πρωί. Όμως τώρα βιάζομαι να φύγω για να μην χάσω το αεροπλάνο. Λυπούμε πάρα πολύ. Λυπούμε λοιπόν, εκφράζω, ε, ζητώ συγγνώμη μάλλον, από την πρόεδρο και από τους και τις συναδέλφους. Ε, θα συνοψίσω εντός ενός λεπτού. Έως τώρα, μάλλον προ δύο ημερών, ε, κατέθεσα το πρώτο σχέδιο, το οποίο συζητήθηκε σε πρώτη συνάντηση των σκιωδών. Ήλθα σε επαφή επίσης με τους αρμοδίους της Επιτροπής για θέματα τα οποία είναι ε, των αρμοδιοτήτων τους. Έχει έρθει τώρα η ώρα της, ε, των τροπολογιών. Έχουμε επιτάπητο σε ένα πρώτο σχέδιο και αναμένω τις τροπολογίες, δεν μπορώ να περισσότερα. Το κείμενο θα είναι σχετικά σύντομο, όλοι συμφωνούμε σε αυτό. και θα αναφέρεται σε ορισμένα κεφαλαιόδη θέματα, διότι βεβαίω μπορεί να γράψει και κανείς 100 σελίδε και να περιλαμβάνει μέσα τα πάντα. Και κάπου χάνεται τότε η ουσία του θέματος. Κάποια από τα κεφαλαιόδη αυτά θέματα είναι το κράτο δικαίου, μετανάστευση, δικαιώματα γυναικών, ελευθερία τύπου και έκφρασης, ρατσισμός, ξενοφοβία και διάφορα είδη διακρίσεων. Στο τέλος του κειμένου αναφέρομαι και για πρώτη φορά σε τέτοιου είδους έγγραφο αναφέρομαι στη σημασία της συμβολής του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, FRA, FRA. Αυτά βρίσκονται όλα βέβαια ακόμα στην φάση της δόμησης. Βρισκόμαστε, ακόμη αν μπορώ να το πω έτσι, στο προ-μαγείρεμα, δηλαδή ετοιμάζουμε τα συστατικά ακόμη, τα οποία θα λάβουν την ε, μορφή τους τις επόμενες ημέρες. Ελπίζω οι συνάδελφοί μου σκιώδεις συζητητές να έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν και άλλες ιδέες στο κείμενο. Ξαναλέω πάλι όμως, σας ζητώ συγγνώμη υποχρεωμένος να αποχωρήσω. Η Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Τερικάμπρας. Τώρα έρχεται η σειρά των σκιωδών εισηγητών για παρεμφάσεις Προσωπικά θα ήθελα να πω μόνο ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ, βρίσκω εξαιρετικό το τμήμα εκείνο της εκθέσεώς σας που αναφέρεται στο κράτος δικαίου. Φρανκ Έγγελ απόν. Ρομπέρτα Μετσόλα επιθυμείτε όχι. Η Ε, είναι βέβαια καμιά φορά δύσκολα τα ονόματα σε άλλε, ε, δυσπρόφατα τα ονόματα σε άλλε γλώσσες. Πράγματι, στη συνάντηση των σκιωδών θέσαμε κάποια θέματα. Τα ξαναλέω και εδώ δημοσία και όσο γίνεται πιο σύντομα για την έκθεση του κ. Τερή Βέβαια, για την μορφή που θα λάβει η έκθεση θα ε, αναφερθούμε στα γεγονότα του 2017. Όμως, δυστυχώς, ορισμένα εκ των θεμάτων είναι και κλασικά και επαναλαμβανόμενα. Πάλι για τον τύπο, είπατε πριν για το κράτος δικαίου, κυρία Πρόεδρε. Θεωρούμε ότι θα είναι χρήσιμο το τμήμα κράτος δικαίου να τονιστεί ιδιαίτερα στο κείμενο και να μπει σε πρωταρχική θέση. Ίσως θα χρειαστεί να δοθεί κάποιος άλλος τίτλος, δηλαδή διακρίσεις με ευρύτερο τρόπο εκεί όπου ε, αναφέρεται σε ξενοφοβία κλπ. Διακρίσεις δηλαδή σε βάρος πληθυσμών μεταξύ αυτών και των αναπήρων. Τα έχουμε πει αυτά στους κοιοδεσίγητες. Θα δούμε που θα καταλήξει η προσπάθεια αυτή. Συμφωνώ με αυτά που λέει ο εισηγητής Τερικάμπρας να είναι δηλαδή μια φιλόδοξη έκθεση, ολοκληρωμένη, είναι όμως δύσκολο και ευαίσθητο το θέμα. Και υπάρχουν τέτοια θέματα τα οποία δεν μπορεί να αποφύγει κανείς. Τώρα, κάποια πράγματα τα οποία η ομάδα μου και εγώ προσωπικά θα τα καταθέσουμε σε τροπολογίες για τα δικαιώματα των γυναικών θα είναι αναγκαίο να προσθεθεί παράγραφος για την ε, γενετήσια παρενόχληση όπως άλλωστε θα χρειαστεί να γίνει παραπομπή και στην ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για το θέμα του κράτους δικαίου. Επανέρχομαι διότι η παράγραφος για την κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να ενισχυθεί. Θα την κάνουμε και πιο περιεκτική. Για ξενοφοβία και εγκλήματα μίσους θεωρούμε αναγκαίο να επιμείνουμε σε κάποιες διακρίσεις που ε, μας φαίνεται ότι δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη, ιδίως για πρόσωπα ε, ομοφιλόφιλα, LGBTI. Σύντομη παρένθεση. Αναφέρονται και κάποιες στατιστικές για διακρίσεις σε βάση της εθνότητας πρέπει να το δούμε αυτό, να φωτιστεί περισσότερο. Για μετανάστευση και άσυλο θα είναι αναγκαίο να γίνουν κάποιες νέες διατυπώσεις και να προσθεθούν κάποια πράγματα και σε νέες κατηγορίες. για θέματα δικαιωμάτων ε, ανηλίκων κλπ. Και αυτά που είπε ο Τζούλιαν Κίνγκ προηγουμένως Θα ξαναδούμε κάποιες διατυπώσεις εκεί και ένα τελευταίο μου φαίνεται σημαντικό να προσθεθεί ένα τμήμα ή και περισσότερα τμήματα για τις ε, πολιτικές χειραγωγήσεις με ψευδή νέα κλπ. Fake news. Αυτά για να παραμείνουμε στα απολύτως αναγκαία στο κείμενο της εκθέσεως. Ευχαριστώ. Εξ όσων κατανοώ, η κυρία Στίβενς αντικαθιστά τον κύριο Γιούρεκ. Ορίστε, έχετε το λόγο, κύριε μου. Dank u wel, voorzitter. Ehm, ik vervang meneer Jurek niet echt, toch niet bij mijn weten. Ik spreek gewoon voor mezelf hier. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει η κυρία Στίβενς ε, δια της διερμηνέως της ε, Φωσεν Κοφάλαλη. Δεν αντικαθιστώ ακριβώς τον κύριο Γιούρεκ, αλλά θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα όσα λέει στην έκθεσή του, ιδίως αναφέρομαι στο άρθρο 21 του κεφαλαίου του, αντίστοιχου κεφαλαίου για θέματα διακρίσεων. Λυπούμε ωστόσο για το γεγονό ότι δεν μιλεί για ανθρώπους με αναπηρίες, διότι ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων αναφέρεται και σε διακρίσεις κατά ανθρώπων με αναπηρίες και τις θεωρεί διακρίσεις. Γιατί αυτή η παράληψη όλες οι χώρες μέλη έχουν κυρώσει το κείμενο αυτό για τα πρόσφατα με αναπηρίες. Διακρίσεις γίνονται ιδίως δε κατά γυναικών και νεαρών κοριτσιών με αναπηρίες όπου προστίθεται και το χαρακτηριστικό του φίλου τους. Όσο έχω τονίσει εγώ ίδια στην έκθεσή μου για το 2016, γυναίκες και νέες κοπέλες με αναπηρίες συχνά υφίστανται βία, ε, καμιά φορά ηθική, καμιά φορά ε, σεξουαλική βία. Γυναίκες και νέα κορίτσια πρέπει να έχουν τις ίσες ευκαιρίες για να μπορούν να παίζουν πλήρως τον ρόλο τους μέσα στην κοινωνία. Παρακαλώ λοιπόν τον εισηγητή και τους κοιόδες εισηγητές για να ληφθούν υπόψη όλες οι μορφές διακρίσεων στην έκθεση και εκεί να, περιληφθεί, να περιληφθούν μάλλον και οι διακρίσεις που γίνονται ε, σε βάρος αναπήρων που είναι σημαντικό. Συχνά μας λησμονούν και εδώ να αποδεικνύεται και πάλι με αφορμή τούτην εδώ την έκθεση. Πρέπει να ενταχθεί μέσα στα πλαίσια μιας στρατηγικής, ευρωπαϊκής στρατηγικής για την πάυση των διακρίσεων σε βάρος αναπήρων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έφτασα με καθυστέρηση αλλά ήμουν σε μια συνεδρίαση για τη Λιβύη. Να ευχαριστήσω καταρχάς τον εισηγητή για τη συνάντηση την οποία είχαμε στην αρχή της εβδομάδας που δείχνει ότι υπάρχει μια πλειοψηφία που θέλει να οδηγήσει σε μια κάποια σύγκληση. Στην αρχή της έκθεσης βέβαια πάντα τα ίδια λέμε και μετά διαπιστώνουμε όταν προχωράμε ότι ο καθένας θέλει να επιβάλλει τα δικά του θέματα. Ο κύριος Έγκελ πέρυσι είχε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια και είχαμε μια επιβλητική σε μέγεθος έκθεση. Σχετικά με τα δημοκρατικά δικαιώματα είναι σαφές ότι πρέπει να τα βάλουμε σε πρώτο επίπεδο γιατί είναι τα θεμέλια της έκθεσής μας. Αξιολογώ θετικά επίσης και τον ρόλο που δίδει ο εισήγητης στην Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Έχω την αίσθηση ότι δεν το κάνουμε συχνά, αλλά μπορούμε να έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για τέτοιου είδους εκθέσεις. Υπάρχουν επίσης δύο στοιχεία τα οποία δεν υπογραμμίζονται αρκετά. Η συνέπεια σε επίπεδο θεμελιωδών δικαιωμάτων της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων που είναι ένα εγκάψιο κατά κάποιο τρόπο θέμα γιατί σε πάρα πολλά θέματα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί ε, έρχεται στην επιφάνεια και δοτίθεται και το σύνεθες ε, αμάλγαμα θα έλεγα η μόνιμη ανάμιξη της νόμιμης ε, μετανάστευσης με την άτυπη μετανάστευση. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, βέβαια κάποιοι μετανάστες οι οποίοι δεν ήταν πραγματικοί μετανάστες και ήταν τρομοκράτες, αλλά είναι σαφές ότι οι αριθμοί είναι ελάχιστοι ε, και φυσικά οι τρομοκρατικές ενέργειες διεξάγονται κατά πλειοψηφία στο ευρωπαϊκό έδαφος από άτομα τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ευρώπη. Βλέπουμε επίσης για την κατάσταση στην Ευρώπη τις τελευταίες μέρες είδαμε ότι παρά την πολύ σημαντική μείωση των αριθμών. Ε, συνεχώς όμως ε, κάποια στοιχεία δείχνουν αυξημένες στατιστικές. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι κατανόητο εδώ. Από τη μία έχουμε πολλά θύματα, από την άλλη έχουμε μείωση του αριθμού. Ε, βλέπουμε επίσης ότι αυξάνεται το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι είναι πραγματικοί πρόσφυγες και οι οποίοι δυστυχώς βρίσκονται σε εξαιρετικά δεινή θέση και πρέπει να μας απασχολήσει. Θα συμφωνήσω και με την κυρία Γκυγιόμ για το θέμα των τεχνικών στατιστικών που στη δική μας χώρα δημιουργεί ένα πρόβλημα. Καλό θα είναι να βρούμε μια ορολογία η οποία θα επιτρέψει τη συνεννόηση. Ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εργαστούμε λοιπόν στα θέματα ρατσισμού, ε, εγκλήματα μίσους ε, και διακρίσεις. Άλλο οι διακρίσεις, άλλο ο ρατσισμός, ξενοφοβία και εγκλήματα μίσους. Γιατί οι διακρίσεις πολλές φορές δεν φτάνουν σε τέτοια επίπεδα και γι' αυτό μπορεί να δημιουργηθεί μια κάποια σύγχυση ανάμεσα στα δύο φαινόμενα. Μένει πάρα πολλή δουλειά που υπάρχει να γίνει. Επίσης τίθεται πολλές φορές και το θέμα της σωρίας ταυτόχρονων διακρίσεων εις βάρος γυναικών, αναπήρων γυναικών, μεταναστριών γυναικών. Υπάρχουν και εδώ πάρα πολλά τα οποία μένει να γίνουν. Δεν έχω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κίνιτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφο Τέρι Κάμπρας για την προσπάθεια την οποία έχει κάνει στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων του 17. Ήταν μια ιδιαίτερα βεβαρημένη χρονιά σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και γι' αυτό χρειάστηκαν πολλαπλές παρεμβάσεις. Όπως είπαν και οι προλαλήσασες, Υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να υπογραμμιστούν ακόμα περισσότερο, όπως το θέμα της ισότητας των φύλων. Δημιουργήθηκαν πέρυσι καταστάσεις θλιβερές ως προς αυτό. Ένα άλλο θέμα, το οποίο κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να τονιστεί, είναι η προστασία των ανηλίκων η οποία αντιμετωπίζεται βέβαια στο κεφάλαιο της μετανάστευσης αλλά με περιορισμένο τρόπο. Έχω την αίσθηση ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να τονιστεί πολύ περισσότερο και να λάβουμε υπόψη μας και άλλες πλευρές όπως η προστασία η νομική, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και τα θέματα της ριζοσπαστικοποίησης των ανηλίκων, της πρόληψης της, θέματα τα οποία περιλαμβάνονται έτσι και αλλιώς και στην ετήσια έκθεση της υπηρεσίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ πολύ. Λόπες Αγουιλάρ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι είναι ε, καταστατική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σαφές στα πλαίσια της αξιολόγησης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αιτήσια βάση στην Ένωση ότι πολλά είναι τα θετικά τα οποία ανακαλύπτουμε. Πέρα από τις πολιτικές μας διαφορές ε, μεταξύ μας και ανάμεσα σε πολιτικές ομάδες οι αρχές αυτές ε, είναι σεβαστές και γίνονται δεκτές από όλους και ό,τι ακούστηκε μέχρι τώρα είναι έγκυρο η σημασία ας πούμε της ισότητας σε ένα τοπίο αυξανόμενων φαινομένων ανισότητας ή το κίνημα μη του τα δικαιώματα των γυναικών που είναι ξανά σε ανωδική πορεία και πολύ σωστό που γίνεται αυτό. Είναι δικαιολογημένο εν πάση περιπτώσει. Γιατί μετά από τόσα χρόνια όπου έχουν καθοριστεί τα πεδία ανισότητας δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά τα οποία μένει ακόμα να γίνουν για τα ισότιμα δικαιώματα των γυναικών. και σε σχέση με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολεως όπως και σε σχέση με τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και τις πρόσφατες επιθέσεις εις βάρος των δικαιωμάτων των γυναικών ακόμα και στο ίδιο το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να συμπληρώσω τα έγκυρα αυτά όπως είπα θέματα με τα θέμα της αντιμετώπισης όλων των μορφών ανισοτήτων και ε, στα πλαίσια όμως των νομικών ρυθμίσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε. Το κράτος δικαίου και αυτό υφίσταται επιθέσεις δυστυχώς στις χώρες μέλη της Ένωσης και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όταν συζητάμε θέματα μετανάστευσης, θέματα ανθρώπων που ζητούν άσυλο, θέματα συνόδευτων ανηλίκων, θέματα μειονοτήτων οι οποίες δικτυακά υφίστανται επιθέσεις και διακρίσεις και το σύνολο όλων αυτών των προβλημάτων αφορά ε, και στους ομόφιλους συμπολίτες μας όπως επίσης και τους αναπήρους. Συνεπώς λοιπόν ανεξαρτήτως των διαφορών τις οποίες μπορούμε να έχουμε και εγώ σαν σοσιαλιστής με τα μέλη των συντηρητικών ας πούμε, της ομάδας των συντηρητικών δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτά τα οποία είπε η Χέλγα Στίβενς για τον ρόλο των γυναικών που συμβολίζουν την κορύφωση ουσιαστικά εις βάρος τους των διακρίσεων. Στην ουσία πρόκειται για μία φάση, σε μία συνεχή διαδικασία. Πρέπει να συνεχίσουμε την πίεση πολέμησης των διακρίσεων γιατί εδώ η έκθεση αυτή παίζει πραγματικά πολύ σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ. Και εγώ λέει η Πρόεδρος να ζητήσω τώρα από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν θέλει να πάρει το λόγο. Να συγχαρώ και εγώ τον κύριο Τέρη Κάμπρας για την έκθεσή του. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομεί τους οποίους μπορούμε να δράσουμε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών μάλλον δικαιωμάτων. Στους έξι τομείς ε, δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε. Νομίζω ότι μερικές φορές ε, η κατάσταση περιγράφεται ίσως λίγο σκοτεινή και δεν αναφέρεται σε κάποια θετικά στοιχεία τα οποία έχουν γίνει για την αντιμετώπιση, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σοβούν στον συγκεκριμένο τομέα. Ας πούμε τα δικαιώματα των γυναικών ήταν κεντρικό σημείο της δραστηριότητάς μας πέρυσι. Αφιερώσαμε και διάφορες συναντήσεις και τα θέματα της μετανάστευσης και των ανηλίκων όπου έχουν γίνει αρκετά θέματα. Επίσης δημιουργήθηκε, όπως ξέρετε, ένα δίκτυο μόνον το θέμα της προστασίας των καταγγελών των δημοσίου συμφέροντος και εκεί έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα. Νομίζω ότι ε, δεν αρκεί να απαριθμούμε αποκλειστικά τα προβλήματα τα οποία πράγματι υπάρχουν, αλλά να, να σημειώσουμε και αυτά τα οποία κάνουμε και είναι αρκετά. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι τροπολογίες ε, πρέπει να κατατεθούν στις 2 μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2018 στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Και περνάμε στο σημείο 10. Colleagues, Συνάδελφοι, το επόμενο σημείο είναι οι δέσμοι για τις ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά δύο μέσα, έναν κανονισμό και μια οδηγία. Όσον αφορά συγκεκριμένη νέα προσέγγιση για τη συγκέντρωση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων. Eurojust και θα αρχίσει να ισχύει το Μάιο και έχει μάλλον αρχίσει να ισχύει από το 2017. Έχουμε δύο οδηγίες για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Ερεύνης. Ε, να σας θυμίσω ότι εκείνη η οδηγία καλύπτει την αμοιβαία αναγνώριση ερευνητικών μέτρων και υιοθετήθηκε μέσω συνένεσης όλων των πολιτικών ομάδων και ο εισηγητής ήταν ο κύριος Νούνο Μέλο. Ε, αυτή η πρόταση τώρα εισάγει καινοτόμα ε, στοιχεία ε, για όσον αφορά το αίτημα για ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία όπως εξοεδαφική εφαρμογή νόμου και εφαρμογή της οδηγίας για την αμοιβαία αναγνώριση σχέση δηλαδή μεταξύ της εκδοτικής αρχής και του παρόχου υπηρεσίας ε, και του εκπροσώπου. Αυτά τα σημεία θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε και φυσικά οι απόψει του εισηγητή θα είναι πολύ βασικές. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. From the commission, yes. Ε, to the commission, to Κομισιόν λοιπόν έχει το λόγο για να μας παρουσιάσει και η κυρία Περνιό και ο κύριος Σρέτερ. Η κυρία Σρέτερ. Καλημέρα σας, ε, καλημέρα κυρία Πρόεδρε. Είμαι η Ιζαμπέλ Περνιόν, είμαι τμηματάρχη στην Τέζε Ζούστο που ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Ε, Είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα αυτό το project γιατί είναι ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό για την Κομισιόν. Γιατί, διότι ανταποκρίνεται σε μια πραγματική ανάγκη των εισαγγελέων. Και όντως ποιο είναι το ιστορικό αυτού του φακέλου. Μας επιτρέπει να θυμίσουμε την σημασία και την, τον επίγοντα χαρακτήρα της υιοθέτηση αυτού του ε, θέματος. Μετά από τις επιθέσεις στο Πατακλάν της 13 Νοεμβρίου του 2015 μας προσέγγισε η εισαγγελία του ε, Παρισιού που μας ζήτησε να βρούμε τρόπο να τους, που θα τους επιτρέπει να έχουν πιο γρήγορα πληροφορίες ε, που χρειάζονται. Όταν λοιπόν ήρθαμε σε επαφή με τους εισαγγελείς στο Παρίσι και πολλά μέλη του της Επιτροπής ε, πήγαν στο Παρίσι. Εμείς ε, στο επίπεδο των υπηρεσιών ε, ε, ε, ε, μιλήσαμε μαζί τους και μας είπαν ότι τα μέσα ποινική συνεργασίας λειτουργούν αλλά δύσκολα και συχνά πολύ αργά και σε επίγουσες περιπτώσεις και όλος ιδιαίτερο στην περίπτωση τρομοκρατικών επιθέσεων είναι σημαντικό οι πληροφορίες να κυκλοφορούν πολύ πιο γρήγορα και άρα από την αρχή αυτό το project το στήριξαν πολλές χώρες. Στη συνέχεια όταν δέχτηκε επιθέσεις και το Βέλγιο δυστυχώς στο Μάλμπεκ και στο αεροδρόμιο οι εισαγγελείς εδώ ήρθαν και εκείνοι να μας πούν ότι χρειάζονται ένα νέο τρόπο ανταλλαγής ε, πληροφοριών. Εξ αρχής λοιπόν πολλές χώρες κινητοποιήθηκαν που γιατί τις, άγγιξε, ή, τις άγγιξαν αυτές οι επιθέσεις ε, αλλά και οι χώρες που είχαν προβλήματα για να έχουν γρήγορα πληροφορίες από τους παρόχους υπηρεσιών. Η Κομισιόν λοιπόν εδώ και δύο χρόνια ήρθε σε επαφές εντατικέ με τους ε, ανθρώπους ε, που χρησιμοποιούν όλα αυτά τα στοιχεία να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες τους ακριβώς, ποιες ήταν οι τι μπορούσε να υλοποιηθεί. Και καταλήξαμε σε αυτές τις δύο προτάσεις που εγκρίθηκαν στις 17 Απριλίου και η Τάνια θα σας παρουσιάσει το περιεχόμενο. Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσω με δύο λόγια για το ποιες είναι οι προτάσεις και ποια είναι τα προβλήματα που προσπαθούμε να καλύψουμε με αυτές τις δύο προτάσεις. Η πρώτο στο σημείο κίνηση είναι ότι τα αποδεικτικά στοιχεία, ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένα δηλαδή που υπάρχουν σε κάποιο format, είτε είναι email, είτε είναι messenger, είτε είναι κάποιο άλλο στοιχείο. Ε, χρειάζονται όλο και περισσότερο για, για τις ε, έρευνες, όχι μόνο για τις κυβερνοέρευνες, αλλά και γιατί αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να αποτελούν κομμάτι οποιοδήποτε ε, είδους έρευνας, για οποιοδήποτε είδους αδικήματος ή εγκλήματος, γιατί όλο ένα και περισσότερο βασιζόμαστε σε αυτές τις υπηρεσίες και που μας προσφέρονται ηλεκτρονικά, χρησιμοποιούμε ε, για να επικοινωνούμε, για να αποθηκεύουμε στοιχεία και το ίδιο κάνουν και οι εγκληματίες. Γι' αυτό και είναι φυσιολογικό ότι η σημασία αυτών των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων αυξάνεται. Ειδικότερο πρόβλημα είναι ότι ε, οι διεθνείς συναλλαγές είναι δύσκολες. Οι πάροχοι των υπηρεσιών Microsoft, Facebook, Google και, και, και μικρότεροι όμως φορείς, ε, πλατφόρμες συχνά ε, παρέχουν αυτές τους τις υπηρεσίες από το εξωτερικό και δεν είναι μόνο ξένες εταιρείες αλλά χρησιμοποιούν και διάφορους τρόπους αποθήκευσης των στοιχείων. Μπορεί ας πούμε μια εταιρεία να είναι εγκαθιδρυμένη σε μια χώρα ενώ η αποθήκευση των δεδομένων της να γίνεται σε μια άλλη χώρα που παρέχει υπηρεσίες και σε άλλες χώρες. για, την, για τις δικαστικές αρχές και για τις αστυνομικές αρχές αυτό είναι πρόβλημα γιατί οι αρμοδιότητές τους σταματούν στα δικά τους σύνορα. Οπότε ε, αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν ε, τα με εργαλεία διεθνούς συνεργασίας και αυτό σε πολλές περιπτώσεις δεν συνδέονται αυτά μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει μια ληστεία στο Βέλγιο και όλα τα στοιχεία της υπόθεσης να, γίνουν, είναι στο Βέλγιο. Δηλαδή, ε, οι δράσεις στο Βέλγιο, οι δράστες Βέλγοι, αλλά οι εγκληματίες να χρησιμοποιήσουν το Messenger του Facebook για να επικοινωνήσουν. Και η αστυνομία θέλω να γνωρίζει ποιος κρύβεται πίσω από κάποιον λογαριασμό. Τότε πρέπει να στραφεί για να ζητήσει τις πληροφορίες στην Ιρλανδία, εάν τα στοιχεία είναι αποθηκευμένα στην Ιρλανδία ή μπορεί να πάει και στη ΣΥΠΑ, να στραφεί στη ΣΥΠΑ για να βρει ποιος είναι ε, πίσω από, αυτήν την, από αυτά τα στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, ε, γι' αυτό τα διεθνή εργαλεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας δεν επαρκούν για να καλύψουν ε, τις ε, προκλήσεις ε, των ερευνών. Τα ηλεκτρονικά στοιχεία είναι στοιχεία τα οποία είναι πολύ εύκολο να διαγραφούν ή και να μετακινηθούν. Και σε μια έρευνα σε μια έρευνα συχνά ξεκινάμε να ζητάμε πληροφορίες ε, για ένα συγκεκριμένο λογαριασμό, μετά ένα δεύτερο βήμα με ποιον επικοινώνησε αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να υπάρξει και ένα τρίτο στάδιο, δηλαδή η, μια έρευνα μπορεί να περάσει πολλά στάδια. Και όπως καταλαβαίνετε ο χρόνος μετράει. Εάν λοιπόν κάθε φορά υπάρχουν καθυστερήσεις, μπορεί να κολλήσει η έρευνα. Η συνεργασία που έχουμε τώρα λοιπόν με τις διαδικασίες αμοιβαία συνεργασίας με τρίτες χώρες και με τις χώρες της Ένωσης, οι διαδικασίες αυτές είναι αρκετά χρονοβόρες και ένα χρόνο μπορεί να πάρουν κατά μέσο όρο οι πληροφορίες να φτάσουν από τις για παράδειγμα. Ε, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι μέγα πρόβλημα όταν πρόκειται για την, ε, τον εντοπισμό ενός υπόπτου. Κάτι άλλο το οποίο στην πράξη έχει αναπτυχθεί είναι ο, θελοντικός, ο μηχανισμός θελοντικής συνεργασίας με τους παρόχους ε, όταν κανείς ψάχνει στοιχεία Αυτή η εθελοντική μορφή συνεργασίας έχει επικρατήσει ως μηχανισμός έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν τα στοιχεία που επιθυμούν οι αρχές. Να σας δώσω κάποια νούμερα. Το 2016 γνωρίζουμε ότι τέσσερις μεγάλοι Αμερικανοί παροχοί έλαβαν 20.000 αιτήματα από τα κράτη-μέλη για τις ηλεκτρονικές, ε, ηλεκτρονικά στοιχεία και αυτό σημαίνει 2.000 ε, ε, αιτήματα συνεργασίας, εθελοντικής συνεργασίας προς τις ΕΠΑ. Το πρόβλημα όμως είναι είναι ότι γενικά ότι δεν, είναι ε, ε, ε, δεν υπάρχει νομική βεβαιότητα όπως θα έπρεπε ούτε για τους, για τις δικαστικές αρχές ούτε για τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται στις διαδικασίες. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε εμείς, τι προτείνουμε και ποια είναι τα κύρια στοιχεία των προτάσεών μας για να καλύψουμε αυτά τα προβλήματα. Το πρώτη μας πρόταση είναι ένας κανονισμός για, την, ε, για το ένταλμα παραγωγής και το ένταλμα διατήρησης μας επιτρέπει να απευθυνθούμε στον πάροχο υπηρεσιών σε κάποιο άλλο κράτος μέλος ε, άμεσα χωρίς να περνάμε από τον μηχανισμό συνεργασίας ε, είναι ένα καινούριο στοιχείο της πρότασής μας που απομακρύνεται από τον ισχύοντα μηχανισμό που λειτουργεί μέχρι στιγμής ότι δηλαδή οι αρχές του κράτους μέλους συμμετέχουν σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ορισμένες υποθέσεις, περιπτώσεις όπου επηρεάζονται τα κράτη-μέλη ή εκεί όπου υπάρχει προφανής ε, κατάχρηση και εκεί ε, όπου χρειάζεται να επιβληθεί η, ε, ε, το ένταλμα επειδή ο πάροχος της υπηρεσίας δεν συμμορφώνεται και δεν συνεργάζεται. Αυτό διότι έπρεπε να βρεθεί ένας γρήγορος μηχανισμός γιατί ο μηχανισμός που υπήρχε δεν επέτρεπε να μειωθούν οι χρόνοι με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό. Δεύτερο θέμα είναι ότι τα κράτη-μέλη είναι ότι Δεν υπάρχει σύνδεση στο κράτος μέλος με την, ε, με την συγκεκριμένη έρευνα. Θα πρέπει να υπάρχει ίσως κάποιος εκπρόσωπος του παρόχου της υπηρεσίας. Θα έπρεπε δηλαδή να χρειάζεται μια αιτιολόγηση για να μπορέσει να συμμετέχει στην έρευνα ο συγκεκριμένο ε, πάροχος. Αυτή είναι η αρχή. Άλλη σημαντική ε, καινοτομία είναι ότι στην προπαρασκευαστική εργασία μας πριν φτάσουμε στην, ε, στην πρόταση συζητήσαμε επί δύο χρόνια Όσον αφορά την αποθήκευση, η αποθήκευση και ο χώρος αυτής ε, αποφασίζεται από τον πάροχο, ε, βασίζεται σε διάφορους παράγοντες. Συχνά είναι άγνωστη η ο χώρος αποθήκευσης, τα, τα στοιχεία μπορεί να κινούνται σε διάφορες ε, αποθηκευτικούς χώρους. Η Google, ας πούμε, έχει ένα τέτοιο pattern που δεν το γνωρίζουμε, ένα τέτοιο σχήμα οι Φιλανδοί ας πούμε, έχουν τεράστια στις αποθηκευτικούς χώρους δεδομένων στη χώρα τους, αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Άλλο σημαντικό θέμα για το μηχανισμό τον οποίο θέλουμε να εισάγουμε είναι ότι εδώ οι πάροχοι των υπηρεσιών λαμβάνουν εντολή, ένταλμα από ένα άλλο κράτος μέλος, το οποίο είναι εγκατεστημένοι το θέμα είναι πώς θα ανταποκριθούν σε, αυτή την, σε αυτό το ένταλμα και πώς οι αρχές θα αντικαταστήσουν η μία την άλλη. Εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών να επιλέγουν αν θα ανταποκριθούν ή όχι, θα πρέπει να ανταποκριθούν από τη στιγμή που τους φτάνει το ένταλμα. Και για τις δικλείδες ασφαλείας που έχουμε φτιάξει, έχουμε δουλέψει πολύ για να ε, βάλουμε ε, δικλίδες για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για το δικαιώματα στη δικαστική διαδικασία, τη δυνατότητα αποθήκευσης των στοιχείων, έχουμε κατόφλια για εγκλήματα, δικήματα, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι μηχανισμοί. Έχουμε ε, ε, η παραδοσιακή αρχή πάντοτε αναμειγνύεται όταν εκδίδεται το ένταλμα παραγωγής, μπορεί να είναι δικαστής, ε, ανάλογα με τα στοιχεία, αναλογικότητα με την ανάγκη των, ε, των απαιτήσεων, την επιταγή. Έχουμε επίσης φτιάξει και αποζημιώσεις για τον άνθρωπο τον, οποίου έχουν χρησιμοποιηθεί τα στοιχεία. Αυτά ξεπερνούν το τι ισχύει σε πολλα κρατημέλη κράτη-μέλη μέχρι στιγμής και τέλος έχουμε φτιάξει και μια ρήτρα για να αντιμετωπίσουμε ε, τις περιπτώσεις σύγκρουσης με νομοθεσίες τρίτων χωρών. Τώρα, για την οδηγία, υποχρέωση για τους παρόχους υπηρεσιών να ορίζουν νομικό εκπρόσωπο. Ε, ε, έτσι ώστε να έχουμε ισότιμο πεδίο και να μπορούν οι αρχές να γνωρίζουν σε ποιον θα απευθυνθούν όταν αναζητούν ηλεκτρονικές, ε, ηλεκτρονικά στοιχεία, καθώς και θα επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών που μπορεί να μην είναι παρόντες στην Ένωση επειδή είναι κάπου αλλού, να έχουν ένα συγκεκριμένο νομικό εκπρόσωπο. Αυτά σύντομα, αυτές σύντομα είναι οι προτάσεις μας πολλά καινοτόμα στοιχεία και πιστεύουμε πως θα αποφέρουν όλα αυτά. Έχουμε δουλέψει πολύ για να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Πιστεύω πως ε, συμπεριλαμβάνονται εδώ πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες. Έχουμε συνεργαστεί με την Προεδρία του Συμβουλίου επικοδομητικά και είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε ε, ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ. Εγώ τώρα, λέει η Πρόεδρος, θα δώσω το λόγο στην κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εξήγησε την επιχειρηματολογία για την πρόταση για ηλεκτρονικά ε, ε, ηλεκτρονικές αποδείξεις. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη συζήτηση για θέματα e-evidence στην Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών. Είχα ωστόσο την ευκαιρία μέχρι τώρα να συζητήσω και με εκπροσώπου της Επιτροπής του Συμβουλίου και μη κρατικέ οργανώσει καθώ και άλλου ενδιαφερομένου. Πολλοί από αυτού μου δήλωσαν ότι οι περισσότεροι φορεί χαίρονται για την ιδέα να εισαχθεί ένα ενιαίο μηχανισμό ποινικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και το γεγονό ότι οι ηλεκτρονικέ αποδείξει θα συνεχίσουν να παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στον χώρο του ποινικού δικαίου, τέτοιο καθεστώ συνεργασία, νέο καθεστώ συνεργασία, ίσω να αποτελεί έναν τρόπο για την αντιμετώπιση υφισταμένων προβλημάτων στη βάση ενό μη διαφανού ε, ε, τρόπου συνεργασίας έως τώρα. Θεωρητικά μπορεί να οδηγήσει σε επιτάχυνση των ποινικών ερευνών. Αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση των αρχών επιβολής του νόμου που αναζητούν δεδομένα, συχνά όμως οι αιτήσει τους δεν οδηγούν ε, πουθενά, είτε διότι υπήρξε καθυστέρηση και τα στοιχεία ή οι αποδείξεις δεν υπάρχουν πλέον, είτε διότι οι αποδείξεις βρίσκονται ε, κατατεθειμένες, αποθηκευμένες δηλαδή, σε service providers αλλού εκτός Ευρώπης και δεν έχουν απολύτως κανένα ενδιαφέρον να βοηθήσουν αυτοί. Ε, αντιλαμβάνομαι επίσης και την ε, απογοήτευση των service providers μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι προσπαθούν ε, λόγω του κατακαιρματισμένου νομικού καθεστώτος και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αιτήσει ε, των αρχών επιβολής του νόμου από διάφορες χώρες μέλη. Τούτων λεχθέντων πάντως, Όλες οι συναντήσεις και τα σχετικά έγγραφα καταλήγουν στο ότι οι προτάσεις όπως έχουν ως τώρα, αντί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη διαφάνεια υπέρ των αρχών επιβολής του νόμου, των providers και των ενδιαφερομένων, ε, οδηγούν μάλλον σε μεγαλύτερη ανασφάλεια δικαίου για όλους τους ενδιαφέρουμενους φορείς και ιδίως ό,τι αφορά τις αρχές των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτή η έλλειψη νομικής ασφάλειας μπορεί να ε, υποσκάψει την επιχειρηματολογία στην οποία βασίζεται η πρόταση δηλαδή την ενίσχυση τη συνεργασία στο ποινικό δίκαιο. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω κάποια από τα βασικά προβλήματα και ανησυχίε σε ό,τι αφορά τι προτάσει. Ο μηχανισμό e-evidence υποτίθεται ότι θα προωθήσει, και αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νέο καθεστώ συνεργασία το οποίο θα επιτρέπει στι νομικέ αρχέ μια χώρα μέλου να ζητεί άμεσα ευθέως αποδείξεις από κάποιον πάροχο υπηρεσιών από άλλη χώρα μέλος ή και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραγωγή και διατήρηση των αποδείξεων δεν εξαρτάται από την έγκριση ε, του ε, αφορομένου προσώπου. Μέχρι τώρα αμοιβαία αναγνώριση σήμαινε μόνο αμοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων μια χώρα μέλου από δικαστικά όργανα άλλη χώρα μέλου. Η νέα πρόταση όμως βγάζει εκτός την δικαστική αρχή της άλλης ε, χώρα μέλου. Παρόλη την, ε, προτάσει συνεργασία συνεργασίας που έχουμε ήδη εγκρίνει, ο ορισμός του ποινικού δικαίου που περιλαμβάνει και τα σχετικά εγκλήματα, προβλεπόμενες ποινές και δικαιώματα, εξακολουθούν να αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των χωρών μελών. Γι' αυτό το λόγο ο ορισμός ή οι ορισμοί εγκλημάτων, ποινών κλπ. έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από χώρας μέλους ή χώρας μέλος. Τότε που είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι οι προτάσεις θα, που έχουμε μπροστά μας θα επιτρέπουν να δίνει εντολή μια δικαστική αρχή χώρας μέλους σε άλλη ε, αρχή χώρας, άλλης, άλλης χώρας μέλους. Μπορεί ωστόσο κάποιε δράσει να θεωρούνται ποινικά δικήματα σε μια χώρα μέλο, όχι όμω σε άλλη. Πολλέ κριτικέ που άκουσα στρέφονται γύρω από την χώρα μέλο όπου βρίσκεται ο service providers. Άλλοι είπαν ότι ιδίω σε ό,τι αφορά ανησυχίες ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων, ασυλίες ή και κρατική ασφάλεια. Μπορεί ε, ε, να μην είναι η χώρα μέλος όπου βρίσκεται ο πάροχο υπηρεσίας, όπου θα είναι αυτή που θα κρίνει εν, τέλος, εν τέλει. Η πρόταση τέλος επιβαρύνει υπερβολικά τον πάροχο υπηρεσιών. Του ζητεί, απαιτεί δηλαδή από αυτόν να ελέγχει την εγκυρότητα και να κρίνει για θέματα εθνικής ασφάλειας κλπ. Όλες, όλοι αυτοί οι έλεγχοι όμως, για, όλα, για όλους αυτούς τους ελέγχους, προβλέπουν οι προτάσεις 10 μόνο ημέρες και σε ορισμένες επίγουσες περιπτώσεις μόνο 6 ώρες. Αυτό οδηγεί σε σημαντική επιβάρυνση των μικρότερων παρόχων υπηρεσιών. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το εξή. Θέλουμε πράγματι στον χώρο του ποινικού δικαίου να οδηγηθούμε σε αποφάσεις ιδιωτών για πολύ θεμελιώδη θέματα όπως για παράδειγμα δικαιώματα στην προσωπική σφαίρα, στην ιδιωτική σφαίρα και μιλώντας για αυτήν εκπλήσωμαι που βλέπω ότι στην πρόταση κανονισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί νέες κατηγορίες δεδομένων που είναι διαφορετικές από αυτές που ήδη έχουν εγκριθεί σε άλλα ε, κοινοτικά νομοθετήματα. Αμφιβάλλω αν κάτι τέτοιο διευκολύνει πραγματικά το έργο των διοκτικών αρχών και των ε, παρόχων υπηρεσιών. Εξάλλου, η πρόταση προβλέπει χαμηλότερα κατόφλια για δύο κατηγορίες όπου υποτίθεται τα δεδομένα είναι λιγότερο ευαίσθητα. Αν εξετάσει κανείς όμως τους ορισμούς, αμφιβάλλει εάν οι κατηγορίες αυτές δεδομένων είναι όντως λιγότερο ευαίσθητες. Εξάλλου, οι τρέχουσες κατηγορίες δεν είναι ξεκάθαρα ορισμένες. Περιλαμβάνουν εν μέρη και τους ίδιους ορισμούς και αυτό επιτρέπει μεγάλη, μεγάλο ε, πεδίο, μεγάλο εύρος ερμηνεών για το τι εντάσσεται σε ποια κατηγορία και αυτό αποδυναμώνει τις εγγύησεις, τις διαδικαστικές εγγύησεις, τις δικονομικές εγγύησεις. Έρχομαι στο επόμενο θέμα των εγγύσεων. Υπό τις παρούσες προτάσεις, σημαντικές δικονομικές εγγύησεις όπως το δικαίωμα ενημέρωσης πληροφόρησης για σχετικό ε, ένομο μέσο ένδικο μέσο δεν είναι εξασφαλισμένη. Και εν ώψη της νέας, του νέου αυτού μηχανισμού οι υποπτοί κατηγορούμενοι θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους σημαντικές δικονομικές εγγύσεις. Τέλος, να μην λησμονούμε ότι ο παρόν μηχανισμός μπορεί να ανοίξει την πηξίδα της Πανδώρας, ενθαρρύνοντας άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισαγάγουν επίσης αμοιβαίε υποχρεώσει για παρόχους υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν δούμε τώρα διάφορε χώρε απανταχού του κόσμου, ορισμένε από τι δικαιοδοσίε αυτέ ίσω να μην ε, σέβονται με τον ίδιο τρόπο ε, θεμελιώδη δικαιώματα και δικονομικέ εγγύσεις όπως εμείς και μάλιστα και μπορεί να πολιτικοποιηθούν ορισμένε υποθέσει. Αν λοιπόν δεχθούμε τέτοιο νέο καθεστώς θα πρέπει να το πράξουμε σωστά και με τις υψηλότερες δυνατές προδιαγραφές ασφαλείας. Όλα αυτά με οδηγούν στο να σκέπτομαι ότι το συγκεκριμένο θέμα χρειάζεται πολλές συζητήσεις, ακόμη πολύ έλεγχο και τώρα ευχαριστώ θα ήθελα να ακούσω από τους κοιόδη συγητάς και συγητρία τι απόψεις έχουν. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, ιδιαίτερα το συνδυάσει κανείς με το EU Privacy. Στην ουσία τα, οι δύο αυτές προτάσεις ε, έχουν κάποια κοινά στοιχεία. Εγώ δεν θα είχα αμφιβολία ή δισταγμούς να δώσω τα προσωπικά μου στοιχεία σε μια, προσωπική, σε μια ιδιωτική επιχείρηση, αλλά Κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτα πάντα δεδομένο όταν πρόκειται για υπηρεσίες κρατικές. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη, είναι σαφές να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ιδιωτικότητας ε, γιατί πράγματι πολλές ε, από αυτές τις επιχειρήσεις δεν δίδουν τις ε, πληροφορίες που πρέπει στις αρμόδιες αρχές με την ταχύτητα που θα έπρεπε. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε τα μέτρα τα οποία θα πάρουμε να είναι τα σωστά. Υπάρχουν κάποιοι τομείς τους οποίους θα πρέπει να υπογραμμίσω. Το χρονοδιάγραμμα, σαν παράδειγμα, εδώ προβλέπετε ότι υπάρχει, θα υπάρχει σε ορισμένες κατεπίουσες περιπτώσεις υποχρέωση απάντηση σε 6 ώρες, αλλιώς σε 10 μέρες. Κοιτάξτε, για μια μεγάλη επιχείρηση αυτό μπορεί να γίνεται, αλλά για μια μικρή επιχείρηση μια μεξικανική πλατφόρμα, δύο άτομα και πηγαίνουν ε, να κοιμηθούν ε, στις 12 ε, δική μας ώρα αλλά προφανώς δεν έχουν απαντήσει κατά τη διάρκεια της περίοδου στα πλαίσια της οποίας είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν πολύ απλά γιατί θα κοιμούνται αλλά ακόμα και μεγάλες επιχειρήσεις ε, όταν ε, λαμβάνουν μια διαταγή δημοσιοποίηση στοιχείων θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι το αίτημα είναι σωστό και πρέπει να δώσουν τις πληροφορίες οι οποίες ζητούνται γιατί αν δώσουν λανθασμένα τις πληροφορίες αυτές είναι κάτι το οποίο στα πλαίσια του GDPR θα μπορούσε να τους κοστίσει μέχρι και το 4% του κύκλου εργασιών τους. Συνεπώς λοιπόν Καταλαβαίνω το κατεπήγον της υπόθεσης, αλλά τα μέτρα τα οποία θα πάρουμε θα πρέπει να είναι λειτουργικά σε ένα σαφές πλαίσιο. Τώρα για αυτά τα οποία είπε η κυρία Σίπελ για τις κατηγορίες των δεδομένων, τις τέσσερις αυτές κατηγορίες, ανησυχώ ιδιαίτερα με τα όρια για πρόσβαση συνδρομητών στα δεδομένα αυτά. Αυτά τα οποία είχα πει στο παρελθόν σε σχέση με τη σημασία της πρότασης αυτής, ιδιαίτερα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, για σοβαρά εγκλήματα όπως δολοφονίες κτλ. Ε, στην Αγγλία ας πούμε έχουν γίνει επανειλημμένα λάθη σε σχέση με τον χαρακτηρισμό υπόπτων οι οποίοι κυκλοφορούν από τη μία είτε ελεύθεροι είτε με ένα δαχτυλίδι παρακολούθησης. Δεν πρέπει λοιπόν να βιαστούμε και γι' αυτό θα ήθελα να μάθω γιατί δεν βάζει χρονικό όριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της σε σχέση με τα δεδομένα των συνδρομητών. Όπως επίσης και την υπερεδαφικότητα, τι ακριβώς γίνεται όταν μία πλατφόρμα βασίζεται σε μία τρίτη χώρα όπου το να δώσει τις πληροφορίες αυτές είναι παράνομο για τους νόμους της συγκεκριμένης χώρας. Οπότε ε, πώς θα μπορέσει το σύστημα αυτό να λειτουργήσει σε διεθνές επίπεδο. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα ήθελα να συζητήσω. Μπας περιπτώσει θα τα συζητήσουμε στο μέλλον. Εγώ υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συνεργαστώ με την κυρία Σίπολ και τους Κιώδης. Η κυρία Ιντβελτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είπε η κυρία Ζίπελ και ο κύριος Ντάλτον, γιατί συμφωνώ σχεδόν με τα πάντα. Έχω αρκετά ερωτηματικά όμως σε σχέση με την πρόταση αυτή και τους λόγους για τους οποίους κατατίθεται. Κοιτάξτε, έχουμε μέσα στη διάθεσή μας, τα οποία από ό,τι μας λένε δεν δουλεύουν πολύ καλά. Μήπως λοιπόν το πρώτο βήμα θα ε, έπρεπε να είναι να διορθώσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία. Δεύτερον, όταν κάθε φορά ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει νέα μέτρα που παραβιάζουν τα δικαιώματα των πολιτών, και εμείς ε, ε, ε, προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα των πολιτών. Κάθε φορά που προτείνουν ένα κατασταλτικό μέτρο θα πρέπει να προτείνουν και μέτρα τα οποία να ενισχύουν την νομική προστασία των πολιτών. Έχουμε μια οδηγία προστασίας δεδομένων, την λεγόμενη αστυνομική οδηγία, η οποία πρώτον δεν έχει εφαρμοστεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών. Μήπως θα έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η εφαρμογή της. Το ότι δεν εφαρμόζεται είναι σοβαρό εμπόδιο στην ανταλλαγή πληροφοριών και δεύτερον είναι μόνο οδηγία. Αυτό αποδυναμώνει την θέση των πολιτών ιδιαίτερα αν αυτές οι λεγόμενες ηλεκτρονικής φύσεως αποδείξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρόπους οι οποία δεν είναι διαθέσιμοι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια λογική εδώ. Αν μπορέσουμε να έχουμε ένα εναρμονισμένο επίπεδο νομικής προστασίας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε πράγματι θα μπορούσε ε, η αστυνομία και οι αρμόδιες υπηρεσίες καταστολής να έχουν άμεση πρόσβαση σε ορισμένα τέτοιου τύπου ιδιωτικά δεδομένα, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει απόλυτα σήμερα. Και δεύτερον, θα συμφωνήσετε μαζί μου, Πρόεδρε, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά για κάποιες χώρες σε σχέση με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης τους. Είδαμε, ας πούμε, ότι μια γυναίκα η οποία εκπροσωπεί μια ΜΚΟ, η οποία ασκεί κριτική στην πολωνική κυβέρνηση, εξεδιώχθη της περιοχής Σέγγεν γιατί υπήρχαν διάφορες κατηγορίες εις βάρος της. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ εύκολο για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές να κάνουν καταχρήσεις σε σχέση με τα δικαιώματα αυτά. Θα πρέπει να καταστήσουμε λοιπόν τα δικαιώματα των ε, πολιτών πραγματικά στεγανά. Μόνο έτσι θα διασώσουμε την, ε, τα, τα συγκεκριμένα αυτά δικαιώματα δύο τελικές παρατηρήσεις. Η μία αφορά τις, ε, τις δικαιοδοσίες και τον ορισμό των δικαιοδοσιών. Νομίζω ότι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις Ηνωμένε Πολιτείε και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι εδώ στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλοι έχουν ισότιμα δικαιώματα. Ε, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη νομική προστασία όπως λέμε στι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα ήθελα να μάθω, και αυτή είναι πολιτική ερώτηση, δεν θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε μέρος στην διαδικασία Microsoft, εναντίον της Microsoft. Και όλοι είχαν πει ότι υπήρχε κάποια σκεπτικό πίσω από αυτό γιατί υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία είχαν ηλεκτρονική προέλευση ε, στην ουσία τι κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα οποία κάνουν και οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ε, ή μα λένε να κάνουμε οι Ηνωμένε Πολιτείε. Αντίθετα, εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε επίπεδο κίνου και μετά νομοθετικές προτάσεις. Θα πρέπει να σταματήσουμε πια να μας επιβάλλουν από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις ανησυχίες και τα μέτρα τα οποία παίρνουμε στον τομέα της ασφάλειας. Θα πρέπει λοιπόν να μην είμαστε <clears throat> απλά υπάκουοι σε ξένες κυβερνήσεις και να παίρνουμε ανεξάρτητα τα μέτρα που πρέπει. Στα πλαίσια λοιπόν της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει ε, να σκεφτούμε με τον πρόεδρο της Επιτροπής να υπάρξει ένα χαρτοφυλάκιο για έναν Ευρωπαίο επίτροπο που θα ασχολείται με τα θέματα της νομικής προστασίας και της προστασίας της ιδιωτικότητας που θα έχει ένα κάποιο θα έλεγα οριζόντιο χαρτοφυλάκιο έτσι ώστε κάθε πρόταση η οποία γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχεται σε σχέση με το σεβασμό της ιδιωτικότητας. Και λόγω της σημασίας που έχουν τα προσωπικά δεδομένα Τώρα μπορούμε να δούμε ότι ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, αγνοεί όλες ε, τις ε, προτάσεις και τις νομοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων σωμάτων όπως και το EDPS. Πρέπει όλα αυτά να προσπαθήσουμε να τα επαναντάξουμε στην λογική μας. Η κυρία Ένστ. Πρόσφατα είχα τονίσει ότι η δική μας πολιτική ομάδα ε, διέπεται από επικοδομητικό πνεύμα. Θα συμπαραταχθώ τώρα με τους Γερμανούς δικηγορικούς συλλόγους οι οποίοι λένε ότι ναι έχουμε κάποια κατανόηση για το γεγονός ότι θέλετε να ε, επιταχύνετε τις διαδικασίες, να τις συντομεύσετε, να είναι ταχύτερα τα πράγματα κτλ. Τα κατανοώ αυτά. Αλλά πόσο, μέχρι πού αυτό είναι το συγκεκριμένο ερώτημα, διότι έχουμε και άλλους μηχανισμούς, όπως ε, την εντολή εκτέλεση έρευνα, investigation order. Ε, πώς οδηγήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στο να θεωρήσει ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να καταθέσει τέτοια πρόταση οδηγίας. Τι πράγματα αξιολόγησε, ποιον ρώτησε, με ποιον διαβουλεύθηκε, από πού προέκυψε αυτή η μεγάλη και επιτακτική ανάγκη να καταθέσει τέτοια πρόταση. Πρώτη ερώτηση αυτή. Πριν δηλαδή να καθιδρύσουμε ένα νέο καθεστώς, ένα νέο μηχανισμό, να δούμε πώς λειτουργούν τα πράγματα που ισχύουν ως τώρα. Λειτουργούν καλά, λιγότερο καλά, αρκετά γρήγορα, λιγότερο γρήγορα. Δεύτερο, η πάροχη υπηρεσιών, αυτή η τρίτη, Μόλι τα ακούω αυτά με πιάνει πονοκέφαλος, διότι δεν ξέρω πώς θα κινηθεί η υπόθεση αυτή, διότι ε, φέρουν μεγάλη ευθύνη αυτοί. Άμα δω τους διαφόρους ε, της ε, Google και συντροφίας, αντιλαμβάνομαι ποια προβλήματα έχουν αυτοί και ποια προβλήματα αποτελούν για μας αυτά. Η ερώτησή μου λοιπόν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η λύση που προτείνεται έχει εξεταστεί. Όλες αυτές οι ευθύνες, άλλωστε η συγγήτρια τα εξήγησε πολύ καλά, η κυρία Ζίπελ δηλαδή. Θεωρείτε ότι είναι πράγματι σωστές οι προτάσεις σας αυτές και ότι πράγματι πρέπει να εκτελέσετε τα όσα σας ζητούν. Και τώρα έχουμε βέβαια και τα διάφορα διαφορετικά νομικά συστήματα στην αγαπημένη μας Ευρωπαϊκή Ένωση με, τη, με τα οποία αντιμετωπίζουμε τόσα προβλήματα. Βλέπουμε άλλα πράγματα στην Πολωνία, άλλα στην Ουγγαρία. Βλέπουμε τελικώ να μην μπορεί να εκδοθεί όπως δεμόν. ευτυχώ λέω εγώ. Ε, είναι πολύ λοιπόν διαφορετικές και οι νομικές αντιλήψεις. Και εκεί πάλι κάπως με πιάνει κέφαλος. όταν βλέπω μια τέτοια ε, ε, ρύθμιση. Έχετε λοιπόν τρόπο να ξεπεράσετε τις δυσκολίες που ε, προκαλούν οι διαφορές των ενόμων συστημάτων. Τώρα, οι δικονομικές εγγύησεις. Πάλι ερχόμαστε εδώ στην προστασία των δεδομένων και λοιπά, τη νέα οδηγία που δεν ξέρουμε κανείς, κανείς δεν ξέρει πώς λειτουργεί. Για μένα το σημαντικό ερώτημα είναι, πάλι απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρείτε ότι τα πράγματα αυτά μπορούν να διασφαλιστούν στην πραγματική πραγματικότητα. Ποιο ελέγχει την τήρηση των δικονομικών εγγύσεων. Για μένα αυτό είναι απολύτως ανοιχτό ερώτημα. Οφείλει λοιπόν κανεί να είναι επιφυλακτικό. Κάθε φορά που πάμε να εισαγάγουμε κάτι τι το νέο, αυτό θα ισχύσει μετά, θα είναι η πραγματικότητα στην ζωή. Θα χρειάζεται λοιπόν να εξετάζουμε κατά πόσο πράγματι πρέπει να επέλθουν κάποιες αλλαγές και αν όντω ο μηχανισμός είναι ορθός. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Μάλιστα, ήσασταν και η τελευταία ομιλήτρια εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Πριν να δώσω τον λόγο πάλι στην κυρία Ζίπελ, θα ρωτήσω πρώτα όμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλει να απαντήσει Μάλιστα, εκπρόσωπος της Επιτροπής. Δεν θα μπορέσω να απαντήσω σε όλα τα σχόλια που έγιναν. Επιλέγω ορισμένα. Πρώτο και σημαντικό. Προτείνουμε τον νέο αυτομηχανισμό και εξήγησα στην αρχή τα προβλήματα και μίλησα και για εθελοντική συνεργασία. Η θέσπιση νομικού πλαισίου δεν σημαίνει ότι δίνεται περισσότερα, περισσότερες εξουσίες στον κατασταλτικούς, κατασταλτικούς μηχανισμούς των ενόμων τάξεων. Και υπάρχει βέβαια και εξασφάλιση των δικαιωμάτων. Δίνει την ευκαιρία δηλαδή να προστατεύονται οι πολίτες. Διαφωνώ λοιπόν με το ότι είναι δίθεν κατασταλτική η διαδικασία αυτή. Μπορούμε να συζητήσουμε βεβαίως και περαιτέρω μέχρι που θα πρέπει να φτάσουν οι δικονομικές εγγύησεις, τα ενδικά μέσα κλπ. Μην λησμονείτε όμως ότι ούτε και η σημερινή κατάσταση εγγυάται όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μιλούμε για πολίτες οι οποίοι επηρεάζονται από ε, διαδικασίες έρευνας και δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι μιλούμε για υπόπτους και κατηγορουμένους, αλλά Οφείλουμε να λάβουμε υπόψη επίσης και τα θύματα των αδίκων πράξεων. Η οδηγία έχει αρχίσει πόλη πριν από ένα χρόνο να εφαρμόζεται, δεν έχει γίνει ακόμα η αξιολόγηση της εφαρμογής της. Γνωρίζουμε για την δικαστική συνεργασία με μηχανισμούς όπως ε, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Συλλήψεως. Να δούμε όμως επίσης ότι Όταν τέθηκε πρώτα-πρώτα το θέμα για τη βελτίωση του τρέχοντος συστήματος, υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλες χώρες μέλη, αλλά όχι από Εγάλο, για να επενδύσουν στο σύστημα, στο μηχανισμό MLA. Και ζήτησαν και γραπτός να υπάρξει εθελοντική συνεργασία με τους παρόχους υπηρεσιών. Υπάρχουν όρια λοιπόν στο τι μπορούμε να κάνουμε. Και γι' αυτό και εμείς επιλέξαμε το περιεχόμενο αυτής της νέας πρότασης και αυτού του νέου μηχανισμού. Στην βάση των όσων ήδη ισχύουν, δηλαδή της εθελοντικής συνεργασίας. Τώρα, για τις κατηγορίες δεδομένων, αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Η διάκριση που κάνουμε ανάμεσα σε, σε ε, συνδρομητές και στην πρόσβαση σε δεδομένα και στα άλλα είδη δεδομένων βασίζονται και στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν έχουμε επινοήσει νέες κατηγορίες δεδομένων. Το μόνο είναι τα access data, τα δεδομένα πρόσβασης. Και μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί περιλαμβάνουμε την αυτή κατηγορία. Υπάρχει πάντως και διάκριση και στην ομολογία του δικαστηρίου και ανάμεσα στα δεδομένα των συνδρομητών και τα δεδομένα των συναλλαγών. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο χρειάζεται να υπάρχει ως αφετηρία των δικαστικών ερευνών για να βρει κανείς ποιος κρύβεται πίσω από ένα συγκεκριμένο λογαριασμό και υπάρχουν δεδομένα τα οποία είναι λιγότερο ευαίσθητα από άλλα. Και επειδή τα ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικές αποδείξεις μπορεί να είναι χρήσιμες για ουδήποτε είδους άδικες πράξεις, όχι μόνο για οργανωσμένο έγκλημα ή για τρομοκρατικές πράξεις κλπ. Πρέπει να αποφευθεί το ενδεχόμενο ατιμορρησίας. Γι' αυτό και προτείναμε εμείς και ένα κατόφλιο για τα subscriber και access data. Και ο ρόλος τώρα των παρόχων υπηρεσιών ήταν και αυτό μια ερώτηση και ένα θέμα στην πρότασή μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Το μέγα πλήθος των ετοιμάτων, των αιτήσεων δηλαδή για την παροχή δεδομένων, απευθύνεται στι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες βεβαίω έχουν και πάρα πολλούς δικηγόρους, οι οποίοι κάνουν σχετικές ε, έρευνες και ελέγχους κάποια δυνατότητα δηλαδή την οποία δεν έχουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ούτε θα ζητήσουμε από τους παρόχους ε, υπηρεσιών να ελέγξουν την εγκυρότητα των αιτήσεων που λαμβάνουν. Βεβαίω την τελική ευθύνη φέρει πάντοτε η δημόσια αρχή και όχι ο παρόχος υπηρεσιών. Θα αρκεστώ σε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει η Πρόεδρος. Θα παρακαλέσω τώρα την Αυστριακή Προεδρία, αν θέλει να κάνει μια σύντομη παρέμβαση. Ένα δύο λεπτά αρκούν. Σας ευχαριστούμε, θα είμαστε σύντομοι. Τα συζητήσαμε τα θέματα αυτά στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Πολλά από τα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν σήμερα από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν γίνει αντικείμενο συζητήσεως ήδη. Βλέπουμε τη σημασία που έχει το συγκεκριμένο θέμα. Αναγνωρίζουμε τη σημασία αυτή και θέλουμε να υπάρξει γρήγορη πρόοδος. Αλλά δεν έχω κάτι άλλο να σας πω σε αυτή τη φάση. Στα πλαίσια αυτής της πολύ δύσκολης υπόθεσης προσπαθούμε και σε επίπεδο αρχών αλλά κυρίως σε επίπεδο πρακτικών λεπτομεριών να βρούμε κάποιες λύσεις. Τους επόμενους μήνες νομίζω θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Η κυρία Ζήπελ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλες και όλους τους ε, σκιώδεις για τις πρώτες αυτές ιδέες που καταθέτουν δεν ακούσαμε δυστυχώς από όλες τις ε, πολιτικές ομάδες σήμερα. Επομένως, θα ε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η πρώτη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, γιατί τότε θα σας ακούσω όλους. Επανέλθουμε σύντομα στην Ευρωπαϊκή ε, Διαταγή Ερευνών, European Investigation Order. Είναι άραγε καλό να αρχίζει κανείς, ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ένα νέο μέτρο όταν μόλις άρχισαν να λειτουργούν οι μηχανισμοί αυτοί και ακόμα δεν έχουμε αξιολόγησή τους. Παρ' όλα αυτά ακούω από όλες και όλους που μίλησαν σήμερα ότι όλοι διατεθειμένοι να συμμετάσχουν στην εργασία, να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του, να συζητήσει τα ανοιχτά θέματα και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κλείσουμε τα κενά που βλέπουμε να υπάρχουν ακόμη. Θα ήθελα με την ευκαιρία να δηλώσω σαφώς ότι το παρόν κοινοβούλιο με όλες τις κοινοβουλευτικές του ομάδες εργάζεται επί όλων των θεμάτων. Το παρόν κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέση για όλα τα θέματα. Συχνά όμως το Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο δεν λαμβάνει αποφάσεις. Είναι απίστευτο το ότι το Συμβούλιο μπλοκάρει τα πράγματα ενώ εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και είμαστε διατεθειμένες να εργαστούμε επί του θέματος. Θα παρακαλέσω το Συμβούλιο να ολοκληρώσει όλα τα εκκρεμή θέματα τα οποία είναι μπλοκαρισμένα ε, για οποιοδήποτε λόγο στο Συμβούλιο. Πολύ ευχαρίστω πάντως θα συναντήσω όλες και όλους τους και να ακούσω τις απόψεις τους, να κάνουμε και επαφές με όλων των ειδών τους εμπειρογνώμονες, ξαναλέω, για να μπορέσουμε να κλείσουμε τα κενά που ε, βλέπουν όλοι στην πρόταση. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεισφορά σας όλων. Δύο και μισή ξαναρχίζουμε.